η απόρριψη της, ε, του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, γάμου, διαζυγίου, κατοικίας και ούτω καθεξής. Εκλογικά δικαιώματα και ε, ποινικό μητρό, πιστοποιητικό για λευκό ποινικό μητρό και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή έντυπα πολύγλωσσα, τα οποία δεν υπάρχουν αυτούσια, αλλά θεωρούνται ως βοήθεια για τη μετάφραση δεν το θέλησε βέβαια αυτό ακριβώς έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τι να κάνουμε. Συζητήσαμε επί μακρόν το ζήτημα της ε, έκδοσης πολύγλωσσων πίστο εντύπων και θελήσαμε το κόστος να μην είναι εξαιρετικά υψηλό. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ε, πιστοποιημένα αντίγραφα ε, για την επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα γίνει μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. Δεν θα είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Έχουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται ατομικά και δημόσια να ενημερώνουν τον πολίτη. Ε, το αποστήλε της Χάγης δεν είναι πλέον απαραίτητο για τα έγγραφα που μπαίνουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού αν αυτό ισχύει σε άλλο κράτος μέλος. Και τέλος έχουμε ρήτρα αναθεώρησης. Δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια έκθεση για να διευρύνει ενδεχομένως το πεδίο εφαρμογής. Για να περιλάβει και τις επιχειρήσεις σε αυτό, αλλά και τα πτυχία και τα πιστοποιητικά δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Και πέντε χρόνια μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει έκθεση όπου θα κάνει την αποτίμηση των θετικών σημείων, των αρνητικών σημείων, των πραγμάτων που δεν δούλεψαν, δεν έφεραν αποτέλεσμα και θα ε, αποφανθεί ενδεχομένω υπέρ τη ή κατά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή αυτού του κανονισμού για να περιλάβει και τι επιχειρήσει και άλλου φορεί. Είναι ε, μία, σε γενικέ γραμμέ κατά την άποψή μου, μία περίπτωση θετική. Ελπίζω ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα βελτιωθεί και θα είναι η συνεργασία καλύτερη από την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα κράτη-μέλη μέχρι σήμερα να έχουν το ένα για το άλλο και έναντι των θεσμικών οργάνων. Ζητώ λοιπόν να εγκρίνετε αυτή τη συμβιβαστική λύση και είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως για κάθε ερώτηση. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Το συζητήσαμε αυτό. Προηγουμένως παρακαλώ να έχετε έτοιμες τις ε, κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι όλοι να ψηφίσετε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Θρίαμβος. 20 υπέρ, ενεστατά. Παρακαλώ κυρία. Μπορείτε να μας πείτε πώς ψηφίσατε. Κατά. Κατά. Το καταγράφουμε. Συγχαρητήρια. Πάμε στο σημείο 12. Πότε θα έχουμε ε, τη συνέχεια, πότε θα πάει αυτό στην Ολομέλεια. Μας μιλάτε για το ποια συνέχεια θα δοθεί ε, στην έκθεση αυτή. το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο σύμφωνα με τη Γραμματεία, λέει ο Πρόεδρος. Να καλωσορίσω μεταξύ ημών τον κύριο Γκίφερ Χόφστατ, διαπραγματευτή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διοργανική Συμφωνία για καλύτερη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, για καλύτερη ε, νομοθετική διαδικασία. Καλωσορίζω και τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Κύριε Φερχόφστατ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου ε, αποστήλατε έτσι ώστε να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Ε, ε βεβαίως μετά από κάθε διαπραγμάτευση ε, αναφέρομαι το ε, Προεδρείο, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, ε, οι βουλευτές και τα μέλη της Επιτροπής σας πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνονται ε, και επίσης και εγώ θεωρώ απαραίτητο να έχω την δικιά σας γνωμοδότηση και άποψη την στιγμή που συνεχίζω τις διαπραγματεύσεις. Ε, έχουμε ομάδες, ομάδες εργασίας εντός των πολιτικών ομάδων ε, και οπωσδήποτε με τον τρόπο αυτό διατηρείται η στενή μας επικοινωνία ε, αλλά και η συνάντηση που έχουμε σήμερα με την, υπηρεσία, με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ξέρετε ξεκίνησαν αμέσως μετά το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή διακοπή οι διαπραγματεύσεις σε δύο επίπεδα. Υπάρχει πρώτον η τεχνική ομάδα με εκπροσώπους από τα τρία θεσμικά όργανα και ε, που συζητούν για τεχνικά θέματα, αλλά υπάρχει και το άλλο πολιτικό επίπεδο ε, υπό τον Υπουργό κύριο Σμιτ, τον κύριο Τίμερ μας πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής και ε, η μόνο των ιδίων που εκπροσωπούμε επομένω την πολιτική άποψη στη συζήτηση των τεχνικών λεπτομεριών. Μέχρι τώρα έχουμε τέσσερις συναντήσεις σε πολιτικό επίπεδο, τελευταία εκ των οποίων έλαβε έλαβε χώρα την 28η Οκτωβρίου ε, και η επόμενη συνάντηση ε, θα λάβει χώρα στη διάρκεια της Ολομελίας τον Νοέμβριο στο Στρασβούργο. Τώρα, αν με ρωτήσετε πού βρισκόμαστε ε, στις διαπραγματεύσεις, θα σας πω κάπου στη μέση, αν όχι ακριβώς στη μέση στη ε, μέση λοιπόν αυτών των διαπραγματεύσεων που βασίζονται σε μια καλή ατμόσφαιρα ε, γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ακριβώς γι' αυτό ευελπιστώ ότι θα έχουμε επιτυχή έκβαση ε, περί το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στον σκοπό της διαπραγμάτευσης και την εντολή η οποία μου δόθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων. Υπάρχουν αρκετά κεφάλαια σε αυτήν την διοργανική συμφωνία και τις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με αυτήν. Θα ήθελα όμως να σας εξηγήσω λίγο σε λεπτομέρεια την ουσία της εργασίας που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το παρελθόν, αλλά να δούμε βέβαια και ποιες είναι οι προσδοκίες μας για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα, μετά από ένα εισηγητικό κεφάλαιο, εισαγωγικό κεφάλαιο, φτάσαμε στο κεφάλαιο 2 των διαπραγματεύσεων που αφορά τον προγραμματισμό. Ε, συζητήσαμε ήδη το κεφάλαιο αυτό του προγραμματισμού και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τελικά μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα μελήματα των τριών θεσμικών οργάνων, ενώ ταυτοχρόνως ε, να διασφαλίζουμε το ε, κύριο μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που είναι ότι οποιαδήποτε και η διοργανική συμφωνία, αυτή η συμφωνία δεν μπορεί ε, να ε, ε, παραβιάσει τη συμφωνία του 2010 μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Ε, αυτή η συμφωνία για καλύτερη νομοθετική ε, διαδικασία δεν αντικαθιστά ή δεν δυναμητίζει ε, το υπάρχον πλαίσιο του 2010. Επομένως θα διασφαλίσουμε στην τελική έκβαση αυτής της διοργανικής συμφωνίας ότι το πλαίσιο συμφωνίας του 2010 θα εξακολουθεί να υπάρχει και να ισχύει μεταξύ του Κοινοβουλίου αφενός και της Κομισιόν αφετέρου. Ε, έχουμε βέβαια και ένα τρίτο εταίρο πλέον, το Συμβούλιο, το, που δεν ήταν εταίρος στη Συμφωνία Πλαίσιο του 2010 και επομένως θα πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση, αλλά παρόλα αυτά είμαστε σε θέση ε, να ε, αναγνωρίσουμε την πλήρη ισχύ και εφαρμογή της συμφωνίας του 2010. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν ε, θα υπάρξουν οι πρόνοιες ε, οι οποίες αφορούν τον πολιετή προγραμματισμό αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό που θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Όπως γνωρίζετε ε, ο πολιετής προγραμματισμός είναι σαφής αφορά τις ε, πολιτικές και τους στόχους που έχουμε για, την, ε, για όλη τη διάρκεια της νομοθετικής περίοδου, ενώ ε, στην άλλη περίπτωση θα έχουμε μόνο τις προβλέψεις για, την, για τον επόμενο χρόνο τα στοιχεία του προγραμματισμού είναι σημαντικά γιατί και τα ετήσια και, ε, και ο ετήσιος και ο πολυετής προγραμματισμός αναφέρονται σε συγκεκριμένα ξεχωριστά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν από τους προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων. Επίσης, το πρώτο κεφάλαιο θα υπάρξουν ε, διατάξεις οι οποίες ε, αφορούν το περιεχόμενο του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν και δεν αναφέρομαι εδώ μονάχα τις, στις κύριες προτάσεις, στις προτάσεις απλούστευσης, ε, στις αποσύρσεις κλπ. αλλά θα αφορά και το βαθμό λεπτομέρειας που θα προβλέπετε σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή ποια είναι η νομική βάση της πρότασης, ε, ε, με ποιου τύπου δράση ε, χρησιμοποιείται, ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έγκρισης της πρότασης κτλ. Επομένως, θα υπάρχει ικανός βαθμός λεπτομερίας όσον αφορά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μόλις σας απαρίθμησα. Επίσης, μελετήσαμε και αναλύσαμε ε, το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2016 ε, και ε, θα δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε βάσει της νέας διαφοροποιημένης προσέγγισης. Ακριβώς δηλαδή βάσει αυτού του κεφαλαίου που θα αφορά την διοργανική συμφωνία και που θα είναι πολύ πιο λεπτομερές. Επίσης, ε, στο κεφάλαιο ε, υποχρεώσεις ε, επιβεβλημένες στην Κομισιόν θα αναφερθούμε στις αποσύρσεις. Η Κομισιόν καλείται να διαβουλευτεί με τους συνομοθέτες και δεν πρέπει εδώ να λησμονούμε ε, και τα αιτήματα για ε, νομοθετικές προτάσεις, ας πούμε, προερχόμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, βάσει του άρθρου 225 των συνθήκων, όπου το αίτημα θα είναι το εξής. Η Κομισιόν να έχει την υποχρέωση να πάντα να ανταποκρίνεται στο έτοιμο του Κοινοβουλίου εντός τριών μηνών, ε, ε, καταδεικνύοντας ε, συγκεκριμένα ε, τι προτίθεται, με ποιο τρόπο προτίθεται να συνεχίσει όσον αφορά την εν λόγω πρόταση. Πάντα στο κεφάλαιο του προγραμματισμού ε, θα, θα θα τροποποιήσουμε λίγο την προσέγγιση προς το Συμβούλιο, δεν το ε, συνηθίζω αυτό, αλλά ε, αναφερόμαστε εδώ σε διμερείς ε, συζητήσεις μεταξύ της Κομισιόν και του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Αυτό ήδη συμβαίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του προηγουμένου βάσει της προηγουμένης συμφωνίας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόνα. Ε, αυτό είναι το γενικότερο θέμα όσον αφορά τον προγραμματισμό και όπως είπα ήδη, Θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, και για να το κάνουμε αυτό ε, θα πρέπει να ε, δούμε με ποιο τρόπο θα τροποποιηθεί ας πούμε η αντιμετώπιση του προγραμματισμένου προγράμματος της Κομισιόν για το 2016. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο αυτής της διοργανικής συμφωνίας που συζητούμε είναι η λεγόμενη better regulation, ε, τα, η καλύτερη νομοθετική διαδικασία και τα καλύτερα εργαλεία για αυτή την νομοθετική διαδικασία που θα βασίζεται πλέον ε, σε εξπόστ αξιολόγηση της νομοθεσίας, ε, δημόσιες διαβουλεύσεις και νέα στοιχεία αξιολόγησης των προτάσεων. Η ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί θα συμπεριλαμβάνει και μία σειρά σημαντικών ε, σημείων που είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολλούς μεταξύ ημών. Αλλά παρόλα αυτά ε, θα αναφερθώ σε αυτά. Πρώτον, η μελέτη αντικτύπου. Αυτό που θα συμπεριληφθεί στη Οργανική Συμφωνία ε, είναι τι θα περιλαμβάνει, τι θα καλύπτει ε, αυτού του είδους ε, η μελέτη αντικτύπου. Μπορεί να είναι για το περιβάλλον, για τα οικονομικά, για, την, ε, για το ανταγωνιστικό περιβάλλον ή αντίκτυπο στο δημοσιονομικό βάρος, ιδίως δε τον αντίκτυπο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, εδαφική και ψηφιακή, συγγνώμη, ψηφιακό και περιφερειακό αντίκτυπο βάσει της αρχής ε, πάντα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας χωρίς να λησμονούμε και θέματα τα οποία άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να μελετώνται και να διαρευνώνται στα πλαίσια ε, της μελέτης αντικτύπου η οποία εξορισμού θα γίνεται από την ε, Κομισιόν για τις νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ε, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς επίσης να δούμε και την αλληλεπίδραση με τις ε, εκτελεστικές ε, και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά αυτό θα το δούμε ξανά και σε άλλο κεφάλαιο, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τις πράξεις αυτές. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να συμφωνήσουμε δηλαδή να αποφασίσουμε για ε, ε, μελέτη ε, αντικτύπου επισημαντικών σημαντικών τροποποιήσεων και βεβαίως η Κομισιόν θα είναι επικεφαλής ας πούμε, αυτών των διαδικασιών και θα υπάρχει και μία Regulatory Scrutiny Board που θα ε, ελέγχει ε, σε βάθος ε, αυτήν την διαδικασία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα είδος ένα είδος ανεξάρτητο ε, πάνελ το οποίο θα είναι εκτός των τριών θεσμικών οργάνων. Ε, αυτό λένε ε, το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Εμείς λέμε όμως ότι η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για αυτές τις μελέτες αντικτύπου. Είναι δικιά τους δουλειά να μελετούν ας πούμε την μελέτη αντικτύπου γιατί μπορεί ας πούμε στη βάση ενός τριμερούς διαλόγου, στα πλαίσια ενός τριμερούς διαλόγου, μέσα στη νύχτα να προκύψει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Η Κομισιόν θα πρέπει να την αναλύσει, θα πρέπει να κάνει τη μελέτη αντικτύπου ε, και την οποία θα πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη μας εάν ε, θέλουμε. Και αν θέλουμε βεβαίως εμείς μπορούμε να κάνουμε και τη δικιά μας μελέτη ε, αντικτύπου μέσω της δυνατότητας την οποία μεταξύ έχουμε δημιουργήσει στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Ε, αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν για την ώρα ε, ε, βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη μελέτη, τις μελέτες αντικτύπου και για μία ακόμα φορά σας λέω ότι δεν λέμε εντάξει θα δημιουργήσουμε έναν εξάρτητο πάνελ, η Κομισιόν θα στείλει δύο ανθρώπους, ε, δύο μέλη, το Κοινοβούλιο θα στείλει άλλα δύο και το Συμβούλιο άλλα τόσα και μετά αυτοί θα μελετήσουν, θα αξιολογήσουν θα εκτιμήσουν την αντικειμενικότητα της μελέτης αντικτύπου. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένας πολιτικός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος. Επίσης, όσον αφορά τα εργαλεία καλύτερης νομοθεσίας, έχουμε το θέμα των δημοσίων διαβουλεύσεων. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις πρέπει να είναι ανοιχτές, πρέπει να είναι διαφανείς και το κύριο είναι ότι αυτές οι ε, ε, διαβούλευση ε, θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα πριν την έγκριση της πρότασης και όχι εκ των υστέρων και όχι μετά. Αρχικά η Κομισιόν είχε αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να διαβουλεύεται με τους εμπλεκόμενους μετά Όταν θα έχει σταλεί λοιπόν το έτοιμα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, γιατί ε, ε, ε, έχουν ήδη οργανωθεί οι πάντες, τα λόμπι χτυπάνε ήδη την πόρτα, την πόρτα μας και την ώρα που η ιδέα αρχική ήταν ότι την ώρα που ξεκινάει η νομοθετική διαβούλευση με εμά να ξεκινήσει και η νομοθετική η, η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Όχι, αυτή η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς θα πρέπει να γίνει πριν και να έχει ολοκληρωθεί όταν θα ξεκινήσει η ε, νομοθετική διαβούλευση. Αυτή η εξπόστα αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι η δημόσια διαβούλευση, η διαβούλευση ε, με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς είναι σημαντική και πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσει η διαδικασία και όχι παράλληλα με τη διαδικασία τη δική μας ε, ε, με τρόπο ώστε να επηρεάζει την ε, ροή της νομοθετικής διαδικασίας. ή εκ των υστέρων εξ αξιολόγηση των εργαλείων και αυτό είναι κάτι σημαντικό θεωρούμε ότι σε αυτό το τμήμα της ε, συμφωνίας ε, θα πρέπει να μελετήσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση ε, των ρητρών της συμφωνίας και κυρίως την λεγόμενη sunset clause. Το τρίτο κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων αφορά τα νομοθετικά εργαλεία. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Η Κομισιόν ξεκίνησε, ξεκινάει με ένα έγγραφο, με ένα, με ένα φάκελο μάλλον, έχει νομική βάση. Όλοι ξεκινούν να ανασκουμπώνονται και να δουλεύουν και στην ε, μέση της ε, διαδικασίας, αυτό μπορεί να συμβεί και σε τριμερή διάλογο, Υπάρχει αίτημα, ας πούμε, από το Συμβούλιο για αλλαγή της νομικής βάσης και το Κοινοβούλιο βγαίνει έξω από την όλη διαδικασία εκδιώκεται. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν τρεις διατάξεις ε, σε αυτό το σημείο, νέες διατάξεις. Γιατί στην παρούσα κατάσταση το μόνο που έχουμε είναι να προσφύγουμε στο δικαστήριο και ενδεχομένως ε, να ελπίζουμε να συνταχθεί με τη δικιά μας άποψη το Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο. Στο μέλλον όμως αυτό που θα συμβαίνει θα είναι το εξή. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξηγεί ε, κάθε νομική βάση και κάθε νομικό εργαλείο, λαμβάνοντας υπόψη ε, της, ε, την διαφορά ανάμεσα σε κανονισμό ή οδηγία. Να προβλέπεται υποχρεωτική ανταλλαγή απόψεων, διάλογος μεταξύ των ε, δύο θεσμικών ε, οργάνων, οποτεδήποτε και εφόσον η Κομισιόν αλλάζει την νομική βάση, ενώ αυτό δεν συμβαίνει τώρα, την αλλάζει και τελείωσε, δεν ε, παίζουμε ρόλο. Και τρίτον, στη συμφωνία θα υπάρχει διέσμευση της Κομισιόν να εκτελεί πλήρως τον ρόλο της μέσω της αξιολόγησης και της διασφάλισης εφαρμογής των συνθήκων ε, και την εφαρμογή της πάγιας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί συνήθως ψάχνουν τα ε, ε, αυτά τα επιχειρήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε την απόρριψη της θέσεως της εκ νέου μελέτης ας πούμε ή από αλλαγής βιαζομικής ε, βάσης. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία νέα εργαλεία τα οποία θα υποχρεώνουν ε, την ε, Κομισιόν για οποιαδήποτε αλλαγή να εφαρμόζει την πάγια νομολογία του δικαστηρίου και τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί και από το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το τρίτο κεφάλαιο ή μάλλον το τέταρτο κεφάλαιο γιατί το τρίτο ε, δεν αποτελεί πραγματικό κεφάλαιο. Το επόμενο κεφάλαιο λοιπόν αφορά τις ε, ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές. Θα υπάρξει σε βάθος συζήτηση. Ε, ο κύριος Άγερ ήταν ο, ο άνθρωπος ε, για τις ε, και εκτελεστικές πράξεις. Ε, εν πάση περιπτώσει εμείς σε, τη, σε αυτό το κεφάλαιο προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια, πετύχουμε κάποια πρόοδο. να σας πω ότι στις διαπραγματεύσεις προέκυψε ότι χρησιμοποιούνται περισσότερο κατεξουσιοδότηση πράξης Ε, και ότι ε, πρέπει ε, και ότι γίνεται μία προετοιμασία με τις, τις Κομισιόν με τους εμπειρογνώμονες που αποστέλλονται στα πλαίσια των ε, του Συμβουλίου και η Κομισιόν θεωρεί ότι ε, ολοκληρώνει τη διαδικασία εκεί και ότι έχει κάνει ε, σωστά τη δουλειά της. Εμείς φρονούμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις συζητήσεις και να μην υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου και τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, ε, στοιχεία συμφωνία ε, όσον αφορά τι κατεξουδότηση και εκτελεστικές πράξεις ε, αφορούν τρία στοιχεία. Πρώτον, μια δέσμευση η οποία θα πρέπει να ληφθεί λαμβάνοντα υπόψη την ευθυγράμμιση με όλου τους φακέλου προ προ-Λισαβόνας. Υπήρχε μια σχετική πρόταση, αλλά απεσήρθη από την Κομισιόν ε, κάτω από το γενικότερο λίμα θέλουμε λιγότερη, καλύτερη νομοθεσία, αλλά τώρα ξαναμπαίνει ε, στο τραπέζι, ίσως όχι με την... Ε, όχι, εμείς δεν θέλουμε υπό την μορφή τροπολογίας ακριβώς, αλλά υπό τη μορφή διαφόρων φακέλων που θα βασίζονται στις θερμοδιότητες κάθε επιτροπή Ας πούμε, για κάθε επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει ένα μίνι ας πούμε για κάθε μεμονωμένη επιτροπή όπως τις γνωρίζουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Επομένως, επανυποβάλλομαι το αίτημα ευθυγράμμισης ε, με τους, ε, τους φακέλους ε, της ευθυγράμμισης με τη Λισαβόνα, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο αυτόν με τον οποίο είχαμε κινηθεί μέχρι τώρα. Δεύτερο στοιχείο για πιθανή συμφωνία όσον αφορά κατεξουσίες και πράξεις είναι ότι τα κράτη ε, ότι, τα, ε, ότι θα δεχτούμε μόνο την ιδέα ότι οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ε, μπορούν να συζητούν βεβαίως στα πλαίσια του Συμβουλίου αλλά ότι και εμείς θα έχουμε πρόσβαση στις συνεδριάσεις και στα έγγραφα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταίο στοιχείο είναι μια ιδέα να δημιουργήσουμε ε, όπως έχουμε κάνει για τις εκτελεστικές πράξεις ε, και για τις κατεξουσιοδότηση ε, πράξεις ένα ίδιο τρόπο αντιμετώπισης. Και μένει μόνο το τελευταίο στοιχείο, δηλαδή ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τα κριτήρια έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε κριτήρια όταν, χρησιμοποιήσουμε, όταν κάνουμε περισσότερο κατεξουδίδες, περισσότερο εκτελεστικές ε, πράξεις για να μην έχουμε κάθε φορά αυτές τις ίδιες διαπραγματεύσεις για κάθε μεμονωμένο φάκελο. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, σημαντική συζήτηση μάλλον. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν χωριστές ε, διαπραγματεύσεις για τα ίδια τα κριτήρια στο μέλλον και επομένως ε, θα είναι κατά κάποιο τρόπο μία ρήτρα η οποία ε, θα αφορά τα κριτήρια ε, τα οποία, τα κριτήρια αποδέσμευσης τα οποία είναι απαραίτητα να εγγραφούν στο προκείμενο θέμα, αλλά αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστή συζητήσεως που θα γίνει στο μέλλον. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την διαφάνεια και τον συντονισμό της νομοθετικής διαδικασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα βάλουμε όλα τα διαφορετικά στοιχεία που αφορούν την διαφάνεια σε ένα και μόνο κεφάλαιο πλέον. Θα συγκεντρωθούν αυτά. Ε, δύο σημεία είναι αυτά τα οποία θα ήθελα κυρίως να υπογραμμίσω. Πρώτον, πρόσβαση στις, ε, ε, στις ε, συνεδριάσεις και τα έγγραφα του Κοινοβουλίου, αυτό είναι, συγγνώμη, του Συμβουλίου, αυτό είναι δύσκολο βεβαίως, γιατί εμείς είμαστε εδώ Κοινοβούλιο, είμαστε ανοιχτοί, έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εργασίας, ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο και ε, δεν πρόκειται το Συμβούλιο να πει «Α, τι θέλετε, πρόσβαση στις ε, συνεδριάσεις μας, άψογα, πολύ ωραία, τις ανοίγουμε σε όλους». Ε, αλλά εμείς έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για, με συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις και καταστάσεις όπου το, το Συμβούλιο δείχνει πραγματικά μεγάλη έλλειψη επιθυμίας και βούλησης να δώσει πληροφορίες στο Κοινοβούλιο. Και επομένως εμείς τους λέμε πέστε μα εσείς, κάντε μας εσείς συμβούλιο μία πρόταση, πέστε μα εσείς συμβούλιο τι είστε διατεθειμένοι να παραχωρήσετε. Ε, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι φυσιολογικό το Κοινοβούλιο να πρέπει να έχει κάποιες πληροφορίες. Επομένως, θέλουμε για πρώτη φορά ε, να υπάρχει τουλάχιστον αναφορά ε, δυνατότητας πρόσβασης του Κοινοβουλίου σε μία σειρά συγκεκριμένων περιπτώσεων ε, στις, στα έγγραφα και τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και αυτό ρητά να το αποδεχθεί το Συμβούλιο. Τουλάχιστον στο πνεύμα της αμοιβαιότητας θα πρέπει να υπάρξει αυτή η πρόσβαση στα έγγραφα. Δεύτερο σημείο, διεθνείς συμφωνίες. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι καταρχήν δεν καλύπτονται οι διεθνείς συμφωνίες ε, μέχρι τώρα, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέον το Κοινοβούλιο έχει πλήρη αρμοδιότητα ε, να ε, εγκρίνει στο τέλος της διαδικασίας την πρόταση του Συμβουλίου και επομένως και επομένως τα πράγματα έχουν ε, αλλάξει. Έχουμε δει ε, ε, Έχουμε δει ας πούμε διάφορες αρνητικές τελικές ψηφοφορίες στην άκτα, σε άλλες περιπτώσεις. Δεν αναφέρομαι στο TTIP γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά εν τέλει εμείς έχουμε ε, μια σημαντική αρμοδιότητα και επομένως ε, η ελλειπής ε, προώθηση πληροφοριών οδηγεί σε αρνητική ψήφο, τελική ψήφο του Κοινοβουλίου και επομένως θα πρέπει να το καταλάβουν το πρόβλημα αυτό γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό, είναι ένα νέο πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα. και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα ε, ε, ε, όπως λέμε ότι πρέπει να έχουμε καλύτερη συμφωνία όσον αφορά την καλύτερη νομοθετική διαδικασία, μια διοργανική συμφωνία όσον αφορά την καλύτερη νομοθετική διαδικασία, θα πρέπει και εδώ να προκύψει μια διοργανική συμφωνία. Να δούμε σε ποιο βαθμό λεπτομέρειας μπορούμε να φτάσουμε σήμερα. Και με ποιο τρόπο και ποιου είδους ε, διευθέτηση μπορεί να γίνει, ποιες πληροφορίες ε, μπορούν και οφείλουν ε, να δίνονται στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μιας διεθνούς συμφωνίας. Αυτό είναι το κεφάλαιο όσον αφορά την διαφάνεια και την, ε, τον συντονισμό, ε, το οποίο κεφάλαιο θα περιλαμβάνει και κάποιες πληροφορίες ε, προς, το, προς τα Εθνικά Κοινοβούλια, βελτίωση αυτής της διαδικασίας δηλαδή, κυρίως μέσω της κοινή ανακοίνωσης των κοινών διαπραγματεύσεων, και την ε, οργάνωση κοινών ε, καταγραφών ε, αυτών των αποφάσεων. Ένα από τα επόμενα κεφάλαια είναι το θέμα της μείωσης του άχθους και ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αλλά δεν καταλήξαμε σε συμπεράσματα με το Συμβούλιο για την μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο και ξέρετε πόσο δύσκολη είναι αυτή η συζήτηση για τους πίνακες ε, συσχετισμού. Αυτό το οποίο λοιπόν προσπαθώ να διαπιστώσω είναι η διάθεση του Συμβουλίου, όχι της Κομισιόν, για το εάν μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο εργαλείο εδώ πέρα. Γιατί έχουμε κολλήσει με τους πίνακες αυτούς ε, συσχετισμού και σύγκρισης, γιατί τους ζητάμε κάθε φορά και μας λένε, τόσο καταλάβατε τι θέλω να πω. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αδιέξοδο. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να βρούμε ένα νέο τρόπο λειτουργίας, ένα εργαλείο στο οποίο θα βάζουμε όλες τις πτυχές της μεταφοράς ε, των οδηγιών κυρίως ε, το χρονοδιάγραμμα το ποσοστό της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ε, που οι Βρετανοί έχουν το υψηλότερο ποσοστό μεταφοράς είναι ενδιαφέρουσα η Βρετανική εμπειρία γιατί κάνουν τη μεταφορά αυτομάτως μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες και μετά αρχίζουν να... τις περικοκλάδες στην υπηρετική Ευρώπη είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε κυβερνήσεις ε, συμμαχικές ε, και το παρακάνουμε με τις ε, περικοκλάδες για να ικανοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ξέρω τι λέω, το έκανα και εγώ επί 9 χρόνια ήμουν στην κυβέρνηση συνασπισμού και ξέρω πως γίνονται τα πράγματα. Είχαμε ακριβώς αυτό το θέμα στα Υπουργικά Συμβούλια. Οπότε θα πρέπει κάπου να ξεκολλήσουμε, να υπάρξει ένα νέο μέσο και τα περιέχει και το χρονοδιάγραμμα και το αποτέλεσμα της μεταφοράς στο Εθνικό Δικαίου και με ποιον τρόπο έγινε η μεταφορά και όλες τις υπόλοιπες ε, περικοκλάδες για να καταλάβουν όλοι με βάση αυτό το μέσο ποιος είναι ο κανονισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οποίο είμαστε εμείς υπεύθυνοι και ποιες είναι οι ρυθμίσεις και πιθανώς υπερβολικές ρυθμίσεις των κρατών μελών γιατί βεβαίως εκμεταλλεύονται την ε, οδηγία. Έχω και πιο προχωρημένα όνειρα αλλά δεν νομίζω πως ε, μπορεί να γίνει κάτι στη συζήτηση. Δηλαδή κάποια στιγμή αν δεν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μία οδηγία να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο κάνει η Βρετανία και να γίνει αυτομάτως. Και η οδηγία θα γίνει άρα κάπως σαν ε, κανονισμός μετά από κάποιους μήνες. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η συζήτηση, η τελική διαπραγμάτευση με αυτή την πρόταση, αλλά θέλω τουλάχιστον να συμφωνήσουμε με την αρχή πως θα υπάρχει ένα νέο εργαλείο που θα αντικαταστήσει αυτούς τους ε, συγκριτικούς πίνακες ε, και θα υπάρχει μια γενική εικόνα του κάθε στοιχείου και της μεταφοράς και του χρονοδιαγράμματος και των προσθέτων πραγμάτων που έχουν μπει. Αυτά για το κεφάλαιο 7. Είπα ούτως ή άλλως πως ε, θέλουμε να προχωρήσουμε με το Κοινοβούλιο από αυτού και νομίζω πως με στηρίζει και η Κομισιόν, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει αυτό. Και τέλος ε, για το επόμενο κεφάλαιο που αφορά την απλοποίηση και την μείωση. Ήδη έχουμε βρει μια γενική περιγραφή του τι θέλουμε να επιτύχουμε, να αποφύγουμε δηλαδή την υπερβολική ρυθμίση και να μειώσουμε το διοικητικό άχθος και αυτό θα μπει ως ορισμός σε ολόκληρο το κείμενο οπότε δεν θα διαπραγματευόμαστε ξανά σε κάθε κεφάλαιο το ποιο είναι ο στόχος αυτής της συμφωνίας και μετά τέλος Θα πούμε ναι, θέμε το χ της 100 ως στόχο μείωσης του διοικητικού άθους ή μήπως είναι καλύτερο αυτό το οποίο προτιμώ εγώ να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα με το οποίο θα υπάρχει μια υποχρεωτική μελέτη στο Κοινοβούλιο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τη μείωση του διοικητικού άχθους γιατί έχω ήδη διαπραγματευτεί 10 φορές νούμερα για τη μείωση του διοικητικού άχθους και μετά δεν γίνεται τίποτα με αυτά τα ωραιότατα νούμερα που διαπραγματευόμαστε. Αυτό το οποίο είναι σημαντικότερο κατά την απόψή μου είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, ένα μηχανισμό ε, έτσι ώστε να μπορούμε να μετράμε αντικειμενικά το τι γίνεται και καθώς έχουμε διάφορες ετήσιες εκθέσεις, ε, π.χ. η έκθεση για την ανάπτυξη, μπορεί να γίνεται μια ετήσια έκθεση για το διοικητικό άχθος στο Κοινοβούλιο, που θα βασίζεται σε μια έκθεση που θα προετοιμάζει η Κομισιόν, οπότε και αυτό είναι επιτάπητος και εδώ πέρα θα ήθελα τις απόψεις σας τι είναι σημαντικότερο είναι τα νούμερα ή είναι να βρούμε ένα νέο μηχανισμό που θα διασφαλίσει πως θα υπάρχει πίεση για να υπάρξει μείωση του διοικητικού άχθους για να έχουμε μια τέτοια αιτήσια έκθεση με τρόπο υποχρεωτικό στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Εκεί είναι λοιπόν οι διαπραγματεύσεις. Όπως είπα είμαστε στο μέσο των διαπραγματεύσεων οπότε την επόμενη φορά θα συζητήσουμε το κείμενο και ναι σας, σας βλέπω κύριε Σάιερ γιατί προσπαθούμε ακριβώς να οριστικοποιήσουμε τα πράγματα στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για τα κεφάλαια 7 και 8 τον Νοέμβριο και όπως σας είπα κύριε Πρόεδρε Είμαι πάντα στην διάθεση της Επιτροπής σας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, για να σας ε, ενημερώσω για τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φερχόφστατ. Τώρα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα ακούσουμε. 5-5 ή δεν ξέρω. Ομαδικά θα δούμε. Κυρία Ρέγνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φερχόφστοτ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε και τις διατυπώσεις σας. Όπως ξέρετε ο διάλογος ξεκίνησε κάπως δύσκολα γιατί πολλά από τα ζητήματα που είπατε αξιολόγηση αντικτύπου, καλύτερες πράξεις, κατεξιοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις ήταν πράγματα στα οποία είχαμε συνεισφέρει. Εγώ ήμουν και στην διάσκεψη των Προέδρων και βλέπω πώς γίνονται με τρόπο σωστό οι πολιτικοί ηγέτες αναλαμβάνουν ευθύνες γιατί στόχος μας είναι να έχουμε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχυρό θεσμικό ρόλο όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και ο πρόεδρος μας μπορεί να πάει και στην διάσκεψη των πρόεδρων και αναμένω και το τι λέει κάθε φορά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, είπατε αρκετά, έχω κάποιες ερωτήσεις. Μιλήσατε για τη δουλειά που κάνετε στο νομικό, στο πλαίσιο της νομικής βάσης. Ε, θα θέλαμε να ακούσουμε λίγα περισσότερα πράγματα γιατί εμείς συνηθίζουμε στην Επιτροπή μας να συζητάμε εις βάθος ε, το ποια νομική βάση θα ε, ισχύσει όταν δεν είναι απολύτως σίγουρο, οπωσδήποτε είναι νομικό. Το ζήτημα είμαστε και βουλευτές βεβαίως και αποφασίζουμε με τρόπο πολιτικό. Οπότε είναι και πολιτικό το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα να δούμε πώς θα έχουν τα ζητήματα. Γιατί υπάρχει το εξή θέμα. λαμβάνεται μία απόφαση και μετά δεσμεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε πώς ε, προγραμματίζεται τα, τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω πως υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν και αν δεν το καλύψουν θα ξαναζητήσω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Γιούτελαντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φερχόφστατ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Και ήθελα να τονίσω και πάλι το ότι η απλοποίηση και η καλύτερη νομοθεσία δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για να οδηγηθούμε σε απορρίθμιση. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, να μην καταλήξουμε σε μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή των κλιματικών στόχων ή την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία. Ακούω κάποια πράγματα που με ανησυχούν. Ούτε πρέπει να εμποδίζει την επίτευξη ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό και για, τις, ε, για τη δικιά σας ε, την δουλειά στις διαπραγματεύσεις για μια διοργανική συμφωνία θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς ως νομοθέτες να κάνουμε κάποιες αναλύσεις και αξιολόγηση αντικτύπου των αποφάσεων μας από τη σκοπιά του φίλου. Θεωρώ πως ως νομοθέτες έχουμε και καθήκον και συμφέρον να δούμε όλα τα σχετικά γεγονότα, να ξέρουμε δηλαδή τι αντίκτυπο έχει μία πρόταση στους πολίτες μας. Αυτό είναι σημαντικό για να αποφευχθεί και το ότι θα προχωράμε σε ένα πεδίο και θα έχουμε ακούσιες συνέπειες που θα οδηγούν σε οπισθοχώρηση σε άλλο. Ισότητα σημαίνει δικαιοσύνη, δημοκρατία και συμμετοχή. Άντρες και γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες να διαμορφώσουν την κοινωνία και τη ζωή τους. Για να γίνει αυτό όμως είναι απαραίτητο εμείς ως νομοθέτες να διασφαλίσουμε ίσα δικαιώματα, ευθύνες ε, και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς ε, της ζωής. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι για να καταλήξουμε, για να ενσωματώσουμε την ισότητα στη λήψη αποφάσεων. Δεν χρειάζεται να σας πείσω γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσω κάποια πράγματα για τις απόψεις σας ε, για την αξιολογησία αντικτύπου με βάση το φύλλο στις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Γιατί νομίζω πως υπάρχει μια ευκαιρία εδώ με την διαδικασία αυτή περί καλύτερης νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ κύριος Καρίμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για το ότι ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που είχαμε, όπου επενείται τους ε, Βρετανούς και εγώ σας ευχαριστώ. Ξεκινάω με αυτό λοιπόν. Αναφέρατε κάτι σημαντικό, μιλήσατε για στατιστικά στοιχεία και πίνακες, αλλά ο εχθρός εδώ πέρα είναι ότι αφενός έχουμε όλες αυτές τις περικοκλάδες ε, και αφενός ε, και αφετέρου δεν χρησιμοποιούνται οι αρμοδιότητες και αυτά τα οποία περιγράφει η οδηγία. Και τίθεται πλέον ζήτημα υπαρξιακό αλλά θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο γιατί υπάρχει αυτή η φράση ε, που λέγεται ότι η Ευρώπη θα υπάρχει μόνο εκεί όπου είναι απαραίτητη. Είναι κάτι το οποίο είναι Ολλανδική ιδέα, αλλά την υιοθετήσαμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα ξεκινήσαμε με αυτό το ζήτημα της αξιολόγησης αντικτύπου. Όπως ξέρετε η Επιτροπή μας ε, παίζει σημαντικό ρόλο, κυρίως με την συνάδελφο την Αγγέλικα Νίμπλερ ε, που φρόντισε να γίνουν τα απαραίτητα βήματα. Το θίξαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά το σκεφτικό αυτό ότι ένα ανεξάρτητο πάνελ από μόνο του είναι απαράδεκτο, είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο και το σκέφτηκα από όταν έγιναν τα τελευταία σας σχόλια και θεωρώ πως ε, να αποδίδεται μεγάλη σημασία στην ικανότητα της Κομισιόν να συντάξει ανεξάρτητες ε, μελέτες ε, αντικτύπου. Ένα από τα παράπονα που ακούω εγώ από τους ενδιαφερόμενους είναι πως συχνά βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία η Κομισιόν κάνει τα πράγματα προθύστερα και χρησιμοποιείται η μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου για να δικαιολογήσει η Κομισιόν την θέση που ήδη έχει. Και από κοινοβουλευτική σκοπιά νομίζω πως έχουμε εδώ πέρα μια μοναδική ευκαιρία να καταλήξουμε σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο μηχανισμό. Και ξέρω πως αυτά τα οποία θέσατε λεπτομερώς ε, την προηγούμενη φορά είπατε δηλαδή το ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα πραγματικά ανεξάρτητο πάνελ γιατί αυτούς τους οποίους διόρισε η Κομισιόν θα θεωρούν πως πρέπει να ακούν την Κομισιόν και η δική μας το ίδιο και του Συμβουλίου το ίδιο. Αλλά μπορούμε νομίζω να το ξανασκεφτούμε. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το δείτε. Μπορούν να δημιουργηθούν μηχανισμοί για να διασφαλίσουμε πως οι διορισμένοι αυτοί δεν θα θεωρούν ότι πρέπει να υπακούν κανένα θεσμικό όργανο αλλά θα πρέπει να σκέφτονται το κοινό καλό. Και σας παρακαλώ λοιπόν να το ξαναδείτε. Ξέρω πως θέλουν να μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι, θα είμαι λοιπόν γρήγορος. Να έρθω τώρα στις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Οπωσδήποτε διαβούλευση, διαφάνεια, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κάποιες πράξεις κατ' εξουσιοδότηση είναι πολύ τεχνικές. παραδείγματο χάρη στην ΕΚΟΝ που κοιτάει κάποια μέτρα επίπεδου 2 σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δουν την ε, διαδικασία αυτή κατά τη διάρκεια της σύνταξης των πράξεων κατεξοδότηση και να μην υπάρχουν ακούσιες συνέπειες. Αυτό θα πω μόνο τις λεπτομέρειες της αφήνωσης σας. Τώρα να αναφερθώ σε κάτι λεπτομερέστερο, κάτι το οποίο το ξέρω καλύτερα, την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Την Ευρώπη μόνο εκεί όπου απαιτείται, όπως λέμε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει αυτός ο έλεγχος στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας και άρα θεωρώ πως είναι σημαντικό η επικουρικότητα να παρακολουθείται σε όλη την νομοθετική διαδικασία. Θα πρέπει δηλαδή, να υπάρχει έλεγχος επικουρικότητας κατά τη διάρκεια και στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι συναδέλφους πως δεν έχει στόχο αυτό να υπονομεύσει το δικαίωμα των βουλευτών να υποβάλουν τροπολογίες. Απλά να σεβόμαστε τις αρχές της επικουρικότητας και της ε, αναλογικότητας ε, και μετά οι ε, βουλευτές θα επιλέξουν πώς θα προχωρήσουν. Ακριβώς για να εφαρμοστεί αυτή η πτυχή του ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει μόνο εκεί όπου είναι απαραίτητη. Παραδείγματος χάρη επικουρικότητα και αναλογικότητα βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η επικουρικότητα θα πρέπει να εξετάζεται στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενδελεχής εξέταση του εάν είναι καλύτερη η δράση στο ευρωπαϊκό από ότι στο εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τρίτον, οι γνωμοδοτήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2011 και 2010, κατά οποίο είναι θετικό αφού σημαίνει πως τα εθνικά κοινοβούλια εμπλέκονται περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να εμπλέξουμε τα εθνικά κοινοβούλια στην ε, δική μας νομοθετική διαδικασία, γιατί έτσι έχουν και ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και αναφερθήκατε και πάλι στα όσα κάνατε και ως Πρωθυπουργό ε, και πολλοί Πρωθυπουργοί παίζουν αυτό το παιχνίδι, κατηγορούν την Ευρώπη για τα μέτρα τα μη δημοφιλή. Πρέπει λοιπόν να τους εμπλέξουμε όχι μόνο μέσω των κυβερνήσεων αλλά και μέσω των κοινοβουλίων. Το Συμβούλιο Μελέτης Αντικτύπου έχει τονίσει το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρικότητα σε πολλές περιπτώσεις οπότε η Κομισιόν πρέπει να το δει αυτό όταν αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για αξιολόγηση αντικτύπου. Πέμπτον, παράταση της περίοδου των 8 εβδομάδων για διαβούλευση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αν το ζητήσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια που θα συμφωνήσουμε με την Κομισιόν με κάποια πολιτική δέσμευση στην οποία θα συμφωνήσουν θεσμικά όργανα και εθνικά κοινοβουλία. Η διαδικασία της κίτρινης κάρτας θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα για τα κοινοβούλια καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου είχαμε δυσκολίες. Αυτό πρέπει να το δούμε. Επιπλέον, πολλά κοινοβούλια έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για ένα μηχανισμό πράσινης κάρτας μέσω της ΚΟΖΑΚ και για να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο και να μπορούν έτσι τα εθνικά κοινοβούλια να κάνουν επικοδομητικές προτάσεις ε, προς την Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν συνάδελφοι πως είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα εθνικά κοινοβούλια να συνεισφέρουν περισσότερο σε μια ε, νωρίτερη φάση της ε, διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ ήθελα να πω και άλλα, αλλά θα τα δώσω κατευθείαν στο γραφείο του Γκί για να μην τρώω το χρόνο της Επιτροπής, γιατί ξέρω πως θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσατε την ευκαιρία. Ευχαριστώ και εγώ εάν συμφωνεί ο κύριος Φερχόφστατ, να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις από τους παριστάμενους και στη συνέχεια να απαντήσει συνολικά ο κύριος Φερχόφστατ. Η κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Γκί Φερχόφστατ ε, για αυτά τα οποία μας είπε. Τα θέματα είναι πολύπλοκα και εύχομαι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, το τέλος του χρόνου πλησιάζει, εγώ απορώ με την αισιοδοξία σας, αλλά τέλος πάντων να αναφερθώ σε κάποιες δήματα. Πρώτον, το θέμα της αξιολόγησης αντικτύπου. Εδώ πέρα χαίρομαι για αυτά τα οποία μας είπατε. Γιατί σε αντίθεση με τον κύριο Καρύμ, εγώ θεωρώ πως ε, είναι υπεύθυνα τα θεσμικά όργανα για τις πράξεις τους και όχι κάποιος άνεξάρτητος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι θεματοφύλακας των συνθήκων, έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας και όταν υποβάλλει μια πρόταση είναι υποχρεωμένη να κάνει αξιολόγηση αντικτύπου και δεν θεωρώ πως ε, πρέπει να παραχωρήσει αυτή την ευθύνη της σε οποιονδήποτε λεγόμενο ανεξάρτητο. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι καλό αυτό το οποίο περιγράψατε σε σχέση και με τον νομοθέτη που πρέπει να έχει την ε, δική του ευθύνη για να κάνει εξήλωση αντικτύπου. Κατόπιν θέσατε ένα ερώτημα για τη μείωση του άχθους. Το ABS το οποίο είπατε, ωραίο αυτό. Κοιτάξτε, Εμένα τα νούμερα δεν μου λένε τίποτα. Σημασία έχει η ποιότητα της νομοθεσίας. Ε, το να λέμε δηλαδή ότι θα πρέπει να διαγράφεται κάποιος νόμος για να δημιουργηθεί ένας άλλος, ε, αυτά είναι μπουρδες. Δεν ε, γίνεται έτσι καλύτερη νομοθεσία. Δεν κάνουμε τίποτα με τα νούμερα. Το ABS όπως το προτείνατε είναι κάτι καλό όσον αφορά όλες αυτές τις περικοκλάδες όπως είπατε που μπαίνουν πάνω στις οδηγίες εδώ πρέπει να προσέξουμε να σκεφτούμε το τι είναι ακριβώς αυτό το φαινόμενο οπωσδήποτε μπορεί να μεταφέρει κανείς αυτολεξή τις οδηγίες αλλά τα κράτη-μέλη έχουν ε, από τις συνθήκες το δικαίωμα να κοιτάξουν τις οδηγίες και να τις προσαρμόσουν ε, στις δικές τους ε, συνθήκες. Το να το λέμε αυτό γραφειοκρατία πραγματικά αμένα με δυσκολεύει. Και δεν είναι και δίκαιο για τα κράτη-μέλη. Τελευταία παρατήρηση. Που προκλήθηκε κάπως από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καρίν για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπωσδήποτε χρειάζεται στενή συνεργασία, αλλά εγώ είμαι υπέρ ενός διαχωρισμού αρμοδιοτήτων και τα, εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δικιά τους τη δουλειά, εμείς έχουμε τη δικιά μας τη δουλειά το να τα, ανακατέψουμε, να τα τώρα όλα αυτά και να μπουν τα εθνικά κοινοβούλια στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία θεωρώ πω είναι λάθος. Έχουν ήδη τη δικιά τους τη δουλειά τα εθνικά κοινοβούλια και είναι αρκετά δύσκολη. Ευχαριστώ, Γκονζάλες Πόνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Η παρέμφασή σας ήταν ειλικρινής, σαφής, εκτεταμένη, γεμάτη λεπτομέρειες. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε λεπτομερέστερα την διαπραγμάτευση υπό εξέλιξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για το επικοδομητικό και συνεργατικό πνεύμα που επιδείξατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Γιατί το σημαντικό είναι να εμπλακούν όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν αρμοδιότητα και να εμπλακούν όλες οι πολιτικές ομάδες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να έχουμε τη δυνατότητα όλοι να παρακολουθήσουμε, να παρακολουθήσουμε τη δουλειά που κάνετε και να ε, γίνουμε κοινωνοί του έργου αυτού. Μπόρεσα λοιπόν με την παρέμβασή σας να διαπιστώσω ότι η πρόοδος ε, υπό τη δική σας κατεύθυνση και διεύθυνση ήταν σημαντική και συνεχίζετε να έχετε τη στήριξη τη στήριξή Η πολιτική μου ομάδα είναι ιδιαίτερο ικανοποιημένη με τις αξιολογήσεις αντικτύπου και τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα, ε, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, διότι όταν έχουμε καλή αξιολόγηση αντικτύπου έχουμε καλύτερη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας και λιγότερη υπερβολική νομοθετική ρύθμιση. Άλλωστε, οι αξιολογήσεις που πρέπει να είναι ανεξάρτητες. Είναι ανεξάρτητες. Αν δεν είναι ανεξάρτητες δεν είναι αξιολογήσεις αντικτύπου. Είναι άλλο πράγμα. Είναι κείμενα επιρρογνωμόνων για τα πεπραγμένα από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να ασκούν κριτική, να είναι ανεξάρτητες για να είναι και χρήσιμες και θα πρέπει να χρησιμεύουν σε όλη τη διάρκεια τη νομοπαρασκευαστικής διαδικασία και όχι μόνο στην αρχή. Στηρίζουμε τη σημασία που δώσατε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και ο κινητήριος μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι οποίες υποφέρουν τα μάλα από, την, από αυτό τον κικαιώνα νομοθετικών ρυθμίσεων ε, που ε, ε, υπάρχει στην Ήπειρό μας και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των εκτονιστέρων αξιολογήσεων αντικτύπου. Άπαξ και τεθεί σε ισχύ νομοθεσία να υπάρξει αξιολόγηση αντικτύπου εκ των υστέρων, για να αξιολογήσουμε τι δεν ε, λειτουργήσε ικανοποιητικά. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβασή σας ως προς τις κατεξουσιοδότηση πράξης και πολύ εμπνευστική θα έλεγα και δεν τολμώ να πω περισσότερα λόγια γιατί έχουμε εδώ άλλους παριστάμενους πιο ε, αρμόδιους όμως ελπίζω επιτέλους να έχουμε ίση μεταχείριση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου να υπάρχει εγγύηση για την ισότητα των όρων και των συνθήκων που διέπουν τα δύο αυτά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα όμως ε, να σας πω κάτι τελευταίο που είναι το εξής. Ε, όλοι θέλουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση καταρχάς να πετύχουμε την ισότιμη μεταχείριση από θεσμικής πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπόν θεσμικών οργάνων και δεύτερον να δώσουμε περισσότερες εγγυήσεις στους Ευρωπαίους πολίτες ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι νόμοι από αυτούς οι οποίοι είναι χρειαζόμενοι και ότι οι διατάξεις είναι ωφέλιμες, είναι χρήσιμες και δεν προσθέτουν και άλλα βάρη στον Ευρωπαίο πολίτη. Και γι' αυτό έχουμε μια σειρά εγγυήσεων, π.χ. της αξιολογήσεις αντικτύπου ή της διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες, τη δυνατότητα ε, συμμετοχής στην νομοθετική διαδικασία από πλευράς του πολίτη και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε δηλαδή μια σειρά τέτοιων εγγυήσεων. Πώς ξέρουμε όμως ότι όλες αυτές οι εγγυήσεις δεν θα μεταφραστούν σε περισσότερη γραφειοκρατία, σε πιο επαχθείς διοικητικές διαδικασίες. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι κάθε φορά που η Ευρώπη προσθέτει εγγυήσεις, το μόνο που προσθέτει τελικά είναι περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερα, περισσότερο, περισσότερη δημόσια διοίκηση. Και εσείς προσωπικά κύριε Φερχόφστατ έχετε ταχθεί, ταχθεί επανειλημμένως υπέρ της μείωσης του, της δημόσιας διοίκησης. Πώς θα τα καταφέρουμε λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ο κύριος Κέστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βεχόστατ. Αυτά τα οποία είπατε. Νομίζω πως συμφωνούμε πως πρέπει να μειωθεί η άχρηστη γραφειοκρατία κυρίως όταν Τραγματικά καταλήγει στο να επιβαρύνει άσκοπα τους ε, πολίτες γιατί έτσι οδηγούμε σε μικρότερη αποδοχή της Ευρώπης. Αλλά παρόλη την ανάγκη μείωση της ε, γραφειοκρατίας ε, θεωρούμε πως η Ευρώπη χρειάζεται κοινωνικούς και δημοκρατικούς κανόνες και όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι πρέπει να προσέξουμε μην καταλήξουμε με το πρόσχημα της μείωσης γραφειοκρατίας να μειώσουμε δικαιώματα εργαζομένων. Παραδείγματο χάρη, ισχύει το ότι οι 24 οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων θα επανεξεταστούν. Είναι νομίζω ουσιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, η προστασία της εργασίας και δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε μείωση των συνθήκων ε, ζωής των εργαζομένων δικαιώματα συναπόφασης, ε, ο βασικός μισθός κτλ. Μιλάμε για καλύτερη ρύθμιση και τελικά θα καταλήξουμε σε μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό αλλά το αναφέρατε και εσείς στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου κατέληξα στο ότι ε, είναι δύσκολο ως βουλευτής εγώ να δω τα διαπραγματικά τα διαπραγματευτικά έγγραφα για την TTIP. Και τι γίνεται τελικά, κυκλοφορούν φήμες για το εάν και κατά πόσον περιέχεται κάτι και μέσα το οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες. Οπότε η διαφάνεια είναι μια σημαντική πτυχή για να καταλήξουμε σε μια σοβαρή συζήτηση η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοχή βεβαίως ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω το οποίο μας απασχολεί στην ε, Γερμανία συνεχώς το ότι δηλαδή στην περιφερειά μου συχνά έχουμε τα έργα με κοινοτική χρηματοδότηση αλλά έρχεται συχνά η καταγγελία, το παράπονο ότι για την εφαρμογή κάποιων έργων υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία για να αποδείξουν πώς χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά. Το έχετε λάβει και αυτό υπόψη. Μήπως θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη ρύθμιση για να διασφαλίσουμε πως αυτά τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κονδύλια να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε σωστά, αλλά να μην έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ, κύριο Σάντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Ως προς την αξιολόγηση αντικτύπου, πιστεύω ότι αυτές οι εκθέσεις είναι μια εξαιρετική ιδέα αλλά θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε ως τρόπο αποφυγής κακών αποφάσεων και όχι ως τρόπο καθυστέρησης και πρόληψης και παρεμπόδισης μάλλον της λήψης καλών αποφάσεων και αν φτιάξουμε ένα κακό ε, σύστημα αξιολόγησης αντικτύπου το δεύτερο ενδεχόμενο θα γίνει πραγματικότητα πολύ φοβούμε και νομίζω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το πρόβλημα κύριε Φερχόφστατ και ε, σας καλώ να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο της ύπαρξης υπερβολικά πολλών μελετών αξιολογήσεων αντικτύπου. Τώρα το θέμα των διαπραγματεύσεων εν μέσω νικτός που οδηγούν σε λήψη κακών αποφάσεων για τις οποίες στη συνέχεια θα χρειάζεται αξιολόγηση αντικτύπου για το κατά πόσο ευνόησαν την κατάσταση ή όχι. Ε, προτείνω μια ρισπροσπαστική λύση να απαγορεύσουμε τους τριμερείς διαλόγους η σοβαρή νομοπαρασκευαστική διαδικασία δεν θα πρέπει να γίνεται από μισοκοιμισμένους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο θέμα εργασιακών συνθήκων για τους πολιτικούς αλλά και για τα μέλη του προσωπικού, του υποστηρικτικού ε, προσωπικού. Ας απαγορεύσουμε λοιπόν τους τριμερείς ε, διαλόγους και νομίζω είναι το καλύτερο για την νομοθετική διαδικασία ως προς τις ρήτρες sunset. Είμαι εξαιρετικός υπέρμαχος τέτοιων ρητρών γιατί καθιστούν πιο εύκολη την αλλαγή των θέσεων όταν κάποιος συνειδητοποιεί ότι η απόφαση που πήρε πριν από χι χρόνια δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. Μπορεί λοιπόν να καταφύγει στη ρήτρα Sunset για να αποφύγει την τελμάτωση. Όμως το Dieselgate, η υπόθεση Volkswagen με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι εάν πρόκειται να έχουμε ρήτρα Sunset τότε θα πρέπει να επιτρέψουμε η οδηγία ή ο κανανισμός να έχει εφαρμοστεί σωστά πριν θέσουμε σε ισχύ τη ρήτρα sunset για την λόγω οδηγία ή τον λόγο κανονισμό. Και τώρα στην περίπτωση του gold plating, της ε, υπερβολικής ε, νομοθετικής διαδικασίας και των ε, ισχυρών μηνυμάτων και της, ε, του στολίσματος της βιτρίνας αν θέλετε νομίζω ότι ο όρος αυτός είναι παραπλιανητικός, έχει αρνητικούς συνειρμούς που δεν ευσταθούν και τέλος ως προς το θέμα της Βρετανίας δεν είμαι και τόσο πεπισμένος όσο είναι ο κύριος Φερχόφστατ και ο κύριος Καρίμ για το ότι ο Βρετανικός τρόπος εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι, αγγίζει την τελειότητα. Έχω την εντύπωση ότι οι Βρετανοί προχωρούν πολύ γρήγορα, εφαρμόζουν τον νόμο κατά γράμμα και μετά συνειδητοποιούν ότι «Οπα, αυτό δεν τα καλή ιδέα σε μας και πρέπει να τα αλλάξουν στη συνέχεια». Και νομίζω ότι αυτό οξύνει τα ευρωσκεπτικιστικά αισθήματα στη χώρα αυτή. Ε, Ευχαρίστω να προσπαθήσετε να με πείσετε ότι σφάλω. Όμως, είναι καλό να εφαρμόζονται τα πράγματα προσεκτικά και να μην ακολουθείτε το γράμμα του νόμου όταν αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ο κύριος Λευγαϊτών, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φεχόφσταντ, ο οποίος ήρθε να μας κάνει ένα πολύ ενδιαφέροντα απολογισμό της διαπραγματικής διαπραγματεύσεων, των διαπραγματεύσεων που έκανε και με πολύ χιούμορ κιόλα. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερο τον Βρετανικό λαό, τον οποίο τιμώ, όμως το να τον παρουσιάσει κανείς ως το καλό ε, μαθητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί θράσος από δική σας πλευράς κύριε Φερχόφστατ. Τώρα, κάτι το, το οποίο μου τράβηξε την προσοχή στην παρέμβασή σας είναι αυτό με την αυτόματη ενσωμάτωση των οδηγιών. Είστε υπέρμαχος και συνήγορος αυτής της ιδέας, ότι δηλαδή αν δεν ενσωματώνεται μια οδηγία μετά το, μετά την, το πέρα συγκεκριμένη προθεσμίας ενσωματώνεται αυτομάτως και αυτοδικαίως στην εθνική νομοθεσία ενός κράτους. Αυτό με, ε, μου έγινε πολλά ερωτηματικά και έχω να σας θέσω καταρχάς τις εξής ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι αυτό συνάδει με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η διαφορά οδηγίας και κανονισμού είναι ότι η οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί από τα κράτη-μέλη ενώ ο κανονισμός άπαξ και εγκρίνεται ισχύει αυτό δικαίως στα κράτη-μέλη γιατί εγκρίνεται από αυτά. Ε, θεωρώ ότι οι προκλήσεις είναι όλο και μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, αλλιώς δεν θα είχα εγώ εκλεγεί και άλλοι σαν και εμένα, θα ήταν πολύ κακή ιδέα να ε, ε, ισχύσει αυτή η αυτόματη και αυτοδίκαιη ενσωμάτωση της οδηγίας μετά το πέρα συγκεκριμένη προθεσμίας, γιατί για άλλη μια φορά τα εθνικά κοινοβούλια τίθενται στο περιθώριο. Ο κύριος Σάιερ, ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερος ε, το ότι ο κύριος Φερχόφστατ ήρθε εδώ για να μας ενημερώσει λεπτομερώς για τις ε, διαβουλεύσεις που είχε, ε, ειδικότερα ως προς τις κατεξουσιοδότηση πράξης που είναι και ένα πρακτικό ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό που μας επιτρέπει να πετύχουμε πολλά πράγματα. Όμως υπάρχει ένα θέμα προγραμματισμού με τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Η συμφωνία πλαίσιο δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ εκτιμώ ιδιαιτέρως. Όμως, κύριε Φερχόφστατ, επιτρέψτε μου να σας πω ότι εκ μέρους του Κοινοβουλίου έχω συμμετάσχει στην κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών και αυτό είναι πολύ σημαντική άσκηση για το Κοινοβούλιο για το θέμα του δικαιώματος ιδίας πρωτοβουλίας ή της έλλειψης δικαιώματος ιδίας πρωτοβουλίας. Κάθε χρόνο πρέπει να προβλέψουμε δηλαδή όλες τις συμβαστικές λύσεις που θα επέλθουν κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, γιατί οι πολιτικές ομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει το περιεχόμενο των θέσεών τους και αυτή η άσκηση είναι ε, πολύ μάταιη και άκαρπη πλάι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ετοιμάζοντας ε, τη δουλειά τη επόμενη χρονιά Και τελικά ε, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό που έγινε πέρσι, που δεν είχαμε ψήφισμα για ε, το φόρτο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ε, δεν έχουν ετοιμαστεί οι συμβαστικέ λύσει. Πώ μπορούμε να ξέρουμε το Δεκέμβριο και να προβλέψουμε για ποια πράγματα θα έχουμε δικαίωμα ίδια πρωτοβουλία για του επόμενου 12 μήνε τη επόμενη χρονιά και να μην μπορούμε για άλλα θα πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο ευέλικτο σύστημα. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ίσως να είναι μια πολύ σημαντική λύση στην πράξη αυτή. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχεδόν σε όλους τους τριμερείς διαλόγους είναι ότι η συζήτηση στρέφεται γύρω από το αν θα κάνουμε κατεξουσιοδότηση πράξη ή κάτι άλλο. Η δική μας Επιτροπή θέλει οριζόντια προσέγγιση σε όλο αυτό το θέμα. Ε, και δεν θέλουμε να έχουμε ε, διαφορετική έκβαση στην Επιτροπή Μεταφορών από την Επιτροπή Οικονομικών, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και ε, δεν έχει καθόλου χαρτιά μοιρασμένα στο, στο χέρι του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το παιχνίδι ως προς την οριζόντια προσέγγιση. Θα σας ακούσουμε, αλλά εμέσως πλην σαφώς και αθεμήτως ενδεχομένως αποδεχόμαστε το θέμα της διαβουλεύσης με τους εμπειρογνώμονες και αυτό το είναι τελείως παράνομο γιατί σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας τέλος η επιτροπολογία, τέλος οι διαβουλεύσεις οι μυστικές με τους εμπειρογνώμονες κτλ. Και όσο δεν υποχωρούμε έναντι του θέματος αυτού από, έναντι από το Συμβούλιο δεν υποχωρούν εκείνοι στα άλλα. Αφού λοιπόν αυτά τα χαρτιά μας μοιράστηκαν πρέπει να τα παίξουμε σωστά και να κερδίσουμε έστω κάτι. Και Η απάντηση που δίνεται είναι ότι ίσως μπορεί να ισχύσουν περισσότερο γενικά κριτήρια και ότι δεν χρειάζεται κάθε διαπραγμάτευση ξεχωριστά να ε, αποφασίσει ότι κάτι θα γίνει με κατεξουσιοδότηση πράξη και το καθεξής που είναι χρονοβόρα διαδικασία, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως με τους διαπραγματευτές εκ μέρους του Κοινοβουλίου, τους συναδέλφους οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι το και το πιο σημαντικό στοιχείο κάθε φορά και το παραχωρούν έναντι ε, ζητημάτων περιεχομένου. Και έρχεται το τελευταίο λεπτό και μας λένε ότι συμφωνούμε σε όλα εκτός από αυτό. Ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και τελικά η εικόνα είναι πολύ ετερογενής, είναι καθόλου οριζόντια και καθόλου ομοιόμορφη ε, ε, σε σχέση με τις διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εάν έχουμε αναγνώριση τη διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες, με δικαιώμα δικαίωμα εποπτείας και εγγύησης, εάν το δεχτούμε αυτό και το παραχωρήσουμε, πρέπει να πάρουμε κάτι από το Συμβούλιο, ότι δεν θα μπλοκάρει δηλαδή τις δικές μας πρωτοβουλίες. Και πρέπει να δεχθεί τη διαφορά μεταξύ των εφαρμοστικών και των κατεξουσιοδότηση πράξεων το Συμβούλιο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός. Είναι δύσκολο αυτό το οικοδόμημα, η δομή η συνθήκη της Λισαβόνας ίσως δεν είναι καλή και βέλτιστη. Είναι καλά αυτά που λέει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως επί χάρτου, γιατί τελικά στην πράξη δύσκολα βρίσκουν εφαρμογή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία κύριε Φερχόφστατ και να ξέρετε ότι ε, θα σας παρακολουθούμε στενά γιατί η Επιτροπή μας έγινε πλέον αρμοδία για την οριζόντια εφαρμογή ε, του περιεχομένου της συνθήκης της Λισαβόνας. Κάτι το οποίο περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαουτάλα και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στα της διαφάνειας λεγόμενα από τον κύριο Φερχόφστατ και χαίρομαι και εκτιμώ ιδιαίτερως ότι για το ότι παλεύεται για το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να έχει πρόσβαση στα έγγραφα και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κάτι το οποίο είναι το τελείως αντίθετο σε σχέση με το πώς δουλεύει το Κοινοβούλιο έναντι του Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να δει όλα τα έγγραφα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε το τέλος του νομοθετικού ε, κύκλου. Οι τριμερείς διάλογοι αυτό είναι. Και νομίζω ότι και ως Επιτροπή και ως Κοινοβουλίο και ως Συμβούλιο έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι και οι πολίτες και το ευρύ κοινό γενικότερα δεν τελούν υποπλήρη σύγχυση σε σχέση με το ποια μπορεί να είναι η ενδυνάμει έκβαση του κάθε, έκβαση του κάθε τριμερούς διαλόγου. Δεν αρκούν αυτά που έχουμε. Θα πρέπει ο τριμερής διάλογος να είναι πολύ πιο προσβάσιμος από το κοινό. Μιλάω για το δικαίωμα της δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα του τριμερούς διαλόγου και με την ιδιότητα μου της εισηγήτριας για τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού 1049 για την πρόσβαση στα έγγραφα από πέρσι θα καταβάλω προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση. Ήδη γίνονται πολλέ προσπάθειες προ αυτή την κατεύθυνση και θέλω να ρωτήσω αν θα με στηρίξετε. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με κάτι που αποτελεί αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένθερμο αίτημα. Και θα ήθελα στο μέλλον να λάβετε υπόψη σας τη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή μας για τις ευρωπαϊκές διοικητικές διαδικασίες και για τη σύνταξη σχετικής νομοθεσίας. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε μια, ένα ενοποιημένο διοικητικό δίκαιο και όχι μια πλειάδα διαφορετικών καταστατικών κωδίκων, δεοντολογίες και το καθεξής. Ε, κάτι το οποίο μπερδεύει τις επιχειρήσεις, μπερδεύει τους πολίτες. Και ευχαρίστω να σας ενημερώσουμε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσάς κύριε Φερχόφστατ, για τη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή μας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας. Είναι μια πρόταση συγκεκριμένη νομοθετική αυτή που έχουμε, που θα βγει στις 28 Ιανουαρίου και την κάνουμε δώρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε να είναι σε θέση να τη δεχτεί. Κύριε Φερχόφστατ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με μία παρατήρηση ε, που βρίσκω πολύ σημαντική, τους τριμερείς διαλόγους και τις νύχτες. Ξέρετε, χωρίς νυχτερινές συνεδριάσεις δεν θα υπάρξουν πολιτικές συμφωνίες. Έχετε δίκιο στην πρότασή σας, αλλά είναι άχρηστη η πρότασή σας. Χρειαζόμαστε πράγματι τις νύχτες και όποιος είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι αυτός που κερδίζει κιόλα. Και γι' αυτό έχουμε και διαπραγματεύσεις και βάλατε εμένα διαπραγματευτή για τη διοργανική συμφωνία γιατί ε, ας πούμε στη βαθιά σιγαλιά της νύχτας εγώ θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση από τον κύριο Σμιτ για παράδειγμα. Φυσική κατάσταση. Όμως, ερχόμενο στις διαφορετικές παρατηρήσεις και στα σχόλια τα διάφορα, καταρχάς για την νομική βάση, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Η ιδέα μας είναι η εξής. Σε κάθε περίπτωση, ποιο είναι το πρώτο βήμα. Η Επιτροπή, η Κομισιόν, εξηγεί γιατί επέλεξε τη χύψη νομική βάση ή νομικό εργαλείο. Δεύτερο βήμα. Εάν το Συμβούλιο ανακοινώσει ή ε, εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής της νομικής βάσης γίνεται αυτή η τριμερή συνάντηση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και συζητείται το ε, λόγο ζήτημα. Και τρίτο στοιχείο, τρίτο βήμα σε αυτή την τριμερή ανταλλαγή απόψεων Απάξει και το Συμβούλιο εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγή τη νομική βάση. Εκεί, από εκεί και πέρα, η Κομισιόν θα έχει δικό ρόλο να διαδραματίσει, γιατί η Κομισιόν είναι που διάλεξε την αρχική νομική βάση. Με βασιζόμενη σε σωστή αξιολόγηση. Φαντάζομαι και η Κάζο, αλλιώ δεν θα την είχε διαλέξει την αρχική νομική βάση και πρέπει η Κομισιό να παίξει το ρόλο τη εκεί, εξηγώντα γιατί θεωρεί ότι είναι κακή ιδέα του Συμβουλίου να αλλάξει την νομική βάση επικαλούμενη τι συνθήκε και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε προβλέψει. Αλλά ας είμαστε ειλικρινεί. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων, πρόκειται για διάλογο. Ελπίζουμε ότι θα πείσουμε με την Επιτροπή το Συμβούλιο να μην πάει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν θέλει ε, το Συμβούλιο να πάει προς αυτή την κατεύθυνση στην πράξη, ο μόνος τρόπος να σταματηθεί είναι να το, να το πάμε στο δικαστήριο. Άρα, είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να, να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κάθε φορά που αλλάζει το Συμβούλιο τη νομική βάση, που θέλει να την τροποποιήσει. Όμως, φυσικά, δεν είναι ένα σύστημα που ε, θα καταστήσει αδύνατο στο Συμβούλιο να αλλάξει τη νομική βάση στο μέλλον. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αναγκαιότητας να προσφύγουμε στο δικαστήριο εάν το Συμβούλιο απλά συνεχίσει να εμένει στην αρχική του ιδέα για τη νομική βάση. Και μάλιστα το Συμβούλιο συνήθως εμένει στη νομική βάση που θέλει το ίδιο, μόνο και μόνο για να ξεφορτωθεί ε, το κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν ε, κρατεοί νομικοί λόγοι για να επιλεγεί η χύψη νομική βάση σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι για να ξεφορτωθεί το ένα από τα δύο σκέλη της νομοθετικής διαδικασίας που είμαστε εμείς. Τώρα, όπως ήδη είπα, Υπάρχει και το θέμα ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με την αξιολόγηση αντικτύπου. Αυτά είναι τα στοιχεία που προβλέπεται να αποτελέσουν ε, τον κορμό της αξιολόγησης αντικτύπου. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και συμφωνώ, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμπεριληφθεί. Τούτων λεχθέντων ως προς την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και τα λεχθέντα υπό τον κύριο Καρίμ, δεν είναι αυτή η διοργανική συμφωνία. Δεν είναι η διοργανική συμφωνία αυτή που θα αλλάξει το μηχανισμό επικουρικότητας και τη ρήτρα επικουρικότητας έτσι όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στη συνθήκη. Ξέρω ποια είναι η διατύπωση της επικουρικότητας στη συνθήκη και ξέρω και πώς συντάχθηκε αυτό. Συντάχθηκε καταρχάς από την ε, συντακτική συνέλευση πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και το Συμβούλιο είχε ε, αναφερθεί πρώτα σε αυτό στη δήλωση του Λάκεν. Και είπαμε ότι αφού είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, ας βρούμε ένα μηχανισμό, είχε υποθεί τότε, να εγγυηθούμε ότι πράγματι εφαρμόζεται η επικουρικότητα. Εξού και προέκυψε στη συνέχεια ο μηχανισμός της επικουρικότητας. Έχει δίκιο ο να να στην ε, στη συνέχεια και να λέει ας την βελτιώσουμε, ναι, θα μπορούσαμε, αλλά δεν είναι συζήτηση, δεν εντάσσεται σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα μπορούσε να είναι αντικείμενο σε μελλοντικέ εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πώ μπορεί κανεί να βελτιώσει το μηχανισμό επικουρικότητα. Και μπορώ να σα πω ότι έχω πράσινη κάρτα ε, υψώνω πράσινη κάρτα στο μηχανισμό αυτό και στην προσθήκη και στην τροποποίηση αυτού του μηχανισμού. Δεν θέλω όμως να αναμειχθούν οι ρόλοι μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Ο κ. Κοφράνη είχε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή τα εθνικά κοινοβούλια ασχολούνται με τις εθνικές αρμοδιότητες και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά θέματα και αν υπάρχει αμφιβολία για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την νομοθετική ότι δηλαδή αυτή η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπαίνει στα χωρικά ύδατα των Εθνικών Κοινοβουλίων, εξού και έχει προκύψει και δημιουργηθεί ο μηχανισμός επικουρικότητας για να διαλευκανθεί το μυστήριο. Όμως δεν μπορεί μια διοργανική συμφωνία να αλλάξει το μηχανισμό επικουρικότητας έτσι όπως έχει προβλεφθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν λειτουργεί το πράγμα με αυτόν τον τρόπο, δεν πάει έτσι. Όμως τέτοιες ιδέες όπως η πράσινη κάρτα που μπορεί να υψώσει το κοινοβούλιο ή όχι, το είπα ήδη στον κύριο Καρίμ. Τέτοιες ιδέες έχουν πέσει στο τραπέζι για την έκθεση σχετική με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εξεταστεί και θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και μετά την έγκρισή της θα ε, πάει και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές του επόμενου χρόνου. Η επικουρικότητα και αναλογικότητα θα είναι βασικά στοιχεία ε, τη αξιολόγηση αντικτύπου ε, στην αρχή αλλά και στο τέλος γιατί πάντοτε έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να προβεί σε μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου. Εάν τελικά στο τέλος της ημέρας ε, μετά το τέλος της νύχτας κατά την οποία έχει διενεργηθεί ένας εξαιρετικός τριμερής διάλογος, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση αντικτύπου fast track με ε, ταχείες διαδικασίες για να δει κατά πόσο έγινε ε, σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας και της αναλλαγικότητας κατά τη διάρκεια του τριμερού αυτού διαλόγου. Δηλαδή πάντοτε μπορεί η Κομισιό να εξετάζει την επικουρικότητα και αναλογικότητα και στην αρχή και στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Έρχομαι τώρα στο θέμα των, του ανεξάρτητου πάνελ. Δεν νομίζω ότι ανεξάρτητο πάνελ είναι τρεις τύποι που ορίζει η Κομισιόν, τρεις τύποι που ορίζει το Συμβούλιο και άλλοι τρεις που ορίζει το Κοινοβούλιο. Αν και δεν θα είναι ισότιμη, θα είναι τρεις από το Κοινοβούλιο, πέντε από το Συμβούλιο, εν πάση τα νούμερα δεν θα είναι ίδια. Ε, ε, και έτσι να είναι όμως, πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την ανεξαρτησία του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει ταυτοχρόνως να αναπτύξουμε τη δική μας δυνατότητα, τη δική μας ικανότητα. Άλλωστε στον οίκο μας το κάνουμε ήδη. Έχουμε περισσότερες από 750 μελέτες, μελέτες αξιολόγησης αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριτίας. Εμείς έχουμε κάνει 35 ως Κοινοβούλιο μελέτες αξιολόγησης αντικτύπου. Το Συμβούλιο έχει κάνει 0. Γιατί όμως, γιατί εκπροσωπεί εθνικές κεντρικές αρχές και διοικήσεις, μπορεί το κάθε κράτος να έχει κάνει εξολόγηση αντικτύπου εσωτερικά, στη δική του εσωτερική δημόσια διοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη δυνατότητα επόπτευσης της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό είναι. Ε, έχουμε ένα Regulatory Scrutiny Board, ένα Συμβούλιο Εποπτείας της Νομοθετικής Διαδικασίας. Και υπάρχει αυτό στη συμφωνία. Και αν υπάρχει αυτό στη συμφωνία, εγώ θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα να ξέρω πώς δουλεύει. Αν είναι εκτός συμφωνίας διοργανικής, γιατί είναι καθήκον και αρμοδιότητα εσωτερική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ε, έχει καλώ να μην μάθω πώ λειτουργεί, γιατί είναι θέμα τη Κομισιόν. Αλλά τότε να μην μπει και στο κείμενο. Αν είναι στο κείμενο τη Διοργανική Συμφωνία, τότε εγώ ω διαπραγματευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να ξέρω πώ δουλεύει αυτό το Συμβούλιο και ποιε είναι οι εγγυήσει για ε, διάφορα θέματα. Μετά από τα σχόλια των συναδέλφων από την Επιτροπή Νομικών ε, Υποθέσεων, π.χ. Εσεί. οι συνάδελφοι μου λέτε ότι θέλετε να βεβαιωθείτε ότι αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου γίνεται με το σωστό τρόπο. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει με ένα ανεξάρτητο πάνελ που θα ε, διευθύνεται από τα τρία θεσμικά όργανα μπορεί να γίνει με το Συμβούλιο Εποπτείας της Κανονιστικής Διαδικασίας που εξετάζει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της αξιολόγησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και άρα στις διαπραγματεύσεις θέλω να μάθω πώς θα δουλεύει, ποιες είναι οι εγγυήσεις. ότι δηλαδή έχει κάνει μια καλή αντικειμενική και ανεξάρτητη δουλειά. Για να μπορέσω να επιστρέψω στα μέλη της δικής σας επιτροπής και στις πολιτικές ομάδες και να πω στον κύριο Καρύμ και στους λοιπούς ε, ότι καλώς ε, ασκήσατε πίεση να υπάρξει ε, ανεξάρτητο πάνελ. Και να καθησυχάσω τις ανησυχίες τους για τη σοβαρότητα αυτού του Συμβουλίου εποπτείας της κανονιστικής διαδικασίας. Αν δεν υπήρχε στο κείμενο της διοργανικής συμφωνίας δεν θα ασχολιόμουν. Αλλά αφού υπάρχει πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα αντικειμενικότητας, ποιότητας της αξιολόγησης αντικτύπου. Επομένως, αυτά είχα να πω, ε, λίγος πολύ για τις ανεξάρτητες αξιολογήσεις, για την επικουρικότητα, την αναλλαγικότητα, το ανεξάρτητο πάνελ, το ενδεχόμενο πράσινης κάρτας στο μέλλον και ούτω καθεξής. Έρχομαι τώρα στα του κύριου Κάουφμαν. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας. Ε, γιατί ε, είσαστε μόνος που είπατε ότι το ABS σύστημα μπορεί να είναι ένα κακό σύστημα. Ε, γιατί, εντάξει, υπάρχουν... Ε, τώρα υπάρχουν άλλα συστήματα, ένα, δύο, τρία, το άλλο έξω, μετά σε λίγο σιγά σιγά θα τα βγάλουμε τα πάντα έξω. Εντάξει, Αυτά τα συστήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά ε, για τις ε, εταιρείε ή για το ίντερνετ, αλλά εμείς είμαστε πολιτικοί και επομένως πρέπει να είμαστε σοβαροί. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε ένα μηχανισμό και πιστεύω ότι μπορούμε εδώ στο σώμα και από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά να, έχουμε, να επιτύχουμε μια συνένεση από αυτού. Έναν ισχυρό μηχανισμό ο οποίος τελικά θα μας οδηγήσει στην σωστή κατεύθυνση, στο σωστό δρόμο. Τώρα ένα έξω, ένα μέσα, 25% δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η προτίμησή μου σαφώς και νομίζω ότι και λαμβάνοντας υπόψη τα, τις, των τελευταίων ημερών πιστεύω ότι υπάρχει συνένεση στο σώμα ε, πέρα από οποιασδήποτε ιδεολογικές διαφορές και προσωπικές προτιμήσει. τίνουμε προ αυτό το σύστημα βεβαίως θα πρέπει να συμφωνήσει, θα πρέπει να πείσουμε ε, την Κομισιόν και το Συμβούλιο, ειδικά το Συμβούλιο όταν πρέπει να ε, δημιουργηθεί έτσι μια ε, υποχρεωτική ετήσια άσκηση στην ε, οποία θα διερευνάτε το κράτος, η κατάσταση της Ένωσης κτλ. Κύριε Γκονσάλες αυτή είναι και η απάντησή μου σε εσά όσον αφορά το πόσα θα ήθελα, πώς θα προτιμούσα να προχωρήσουμε. Ε, νομίζω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο για τη μείωση του βάρους και θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε να το προχωρήσουμε αυτό. Είπα ήδη όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες ότι στις διεθνείς συμφωνίες θα προσπαθήσουμε να ανακοινώσουμε μια ξεχωριστή κίνηση διαπραγματεύσεων για, το, για τις διεθνείς συμφωνίες IIA. Θα είναι ένα είδος ραντεβού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, είναι το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κείμενο. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε ολόκληρο το σύστημα ε, σε αυτήν την ε, ε, IIA. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο σε επόμενες IIA. Διοργανικές συμφωνίες. Επίσης ε, θεωρώ ότι το ζήτημα δεν είναι μονάχα ε, θέμα κανονισμού, είναι θέμα ε, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν και οι δημόσιοι λειτουργοί. Δηλαδή, α, okay, τώρα έχω καλύτερη νομοθεσία, έχω καλύτερη αντιμετώπιση. Όχι, θα πρέπει και η ίδια η, δική, η διοίκηση να προσαρμοστεί, αλλά νομίζω ότι αυτό ούτως ή άλλως καλύπτεται πλήρως από τούτη τη διοργανική συμφωνία. Τώρα το gold plating. Εγώ δεν αναφέρομαι στο gold plating, εγώ αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία ε, σχετίζονται με την ε, εφαρμογή και μεταβίβαση της οδηγίας που δεν εμπίπτουν βέβαια στο πεδίο εφαρμογή οδηγία. Γιατί οτιδήποτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή οδηγία δεν με προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται το κάθε κείμενο είναι πλήρης αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών, αλλά να δούμε εάν σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν είναι αυτό το gold plating. Είναι κάτι που έχω δει πάρα πολλές φορές, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Όταν ε, ήμουν εγώ επικεφαλής ε, του Συμβουλίου των Υπουργών, ότι δηλαδή υπήρχε μία τάση να μπαίνουν μέσα στο νομοθέτημα στοιχεία τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το πεδίο εφαρμογής ε, του νομοθετήματος ε, και μου λέγανε ναι αλλά ξέρετε υπάρχει αυτή η διασύνδεση, υπάρχει αυτό το... Ε, αυτό για μένα είναι το gold plating, αυτό που ονομάζω gold plating. Ε, και πιστεύω ότι κατά αυτή την έννοια θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα, ε, ένα πολύ, να είμαστε πολύ προσεκτικοί κυρίως και όσον αφορά το, τους πίνακες συσχετισμών και αυτό έχει ένα πολύ ωραίο όνομα το ότο που αφορά ε, οτιδήποτε σχετίζεται με την, ε, ε, με τα, με την εφαρμογή της οδηγίας από κράτη-μέλη αλλά που δεν έχουν καμία και που δεν έχει καμία σχέση με το πεδίο εφαρμογής. Γιατί πρόκειται δηλαδή για κάτι το οποίο δεν αφορά καθόλου αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά με μονομένες αποφάσεις των κρατών μελών. Κύριε Λεμπρετών, να σας απαντήσω. Η ιδέα ότι κάποια στιγμή μια οδηγία γίνεται κανονισμός, δεν μπορεί να γίνει έτσι παρά μονάχα εάν ήδη έχει προβληθεί η απόφαση αυτή τη στιγμή της οδηγίας. Δηλαδή να πούμε ότι αυτή έχουμε μια οδηγία, αυτή η οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί ας πούμε σε 12 μήνες και αν αυτό δεν ισχύσει τότε αυτόματα η οδηγία θα γίνει κανονισμός. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί ήδη από την νομοθετούσα αρχή δεν μπορεί να είναι ένα αυτόματο γραφειοκρατικό σύστημα. Αυτό, αλλά σας το λέω ε, εξ αρχής ότι δεν ε, πρόκειται να γίνει αποδεκτό αυτό. Εγώ το λέω έτσι ώστε τελικά να καταλήξουμε σε ένα σύστημα ε, μέσα στο οποίο με καλύτερο τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε ε, την εφαρμογή των κειμένων από πλευρά κρατών μελών, έτσι ώστε να είμαστε έντιμοι απέναντι στους πολίτες. Ε, ε, η εντιμότητα αυτού του είδους μας λέει ότι αυτό που είπε ο κ. Καρίν και άλλοι να είμαστε καθαροί γιατί πολύ συχνά σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιούν την Ευρώπη σαν μπαμπούλα, ενώ τα περισσότερα από αυτά που αναφέρονται στην εφαρμογή της οδηγίας δεν έχουν καμία σχέση με την οδηγία αυτή καθεαυτή. Και δεν είναι οι Βρυξέλλες που εφαρμόζουν, είναι το Παρίσι, είναι το Λονδίνο, είναι το Βερολίνο, είναι δηλαδή η κάθε χώρα μέλος. Και ούτω ή άλλω στι Βρυξέλλε, έτσι κι αλλιώ είναι υπεύθυνε οι Βρυξέλλε. Εδώ είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορούμε να το λέμε πάρα πολύ ωραία. Φταίνε οι Βρυξέλλε. Και τρέχα γύρευε μετά. Πολύ ωραία. Και κάτι άλλο μάλλον. Όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ε, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, όσον αφορά το κεφάλαιο της διαφάνειας δηλαδή. Ξέρουμε ότι και η ε, διαμεσολαβητής, η ombudswoman, έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό της διαφάνειας των τριμερών διαλόγων. Ωστόσο νομίζω ότι δεν είναι θέμα που ο Ομπουτσμάν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, πρέπει να λύσει. Εμείς πρέπει να το λύσουμε. Εμείς ε, οι ασκούντες στην νομοθετική διαδικασία. και μάλιστα σε μια επιστολή προς την ε, Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια και ε, προς τον ε, κύριο Σούλτς ακριβώς αυτό έχουμε αναφέρει. Ενστερνίζομαι λοιπόν την παρατήρησή σας για τον τριμερή διάλογο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, έχω κανένα θετικό στοιχείο ή κανένα στοιχείο πρόοδου να σας ε, αναφέρω, αλλά οπωσδήποτε ε, το σημειώνω και το λαμβάνω υπόψη μου επί τη βάση και της επιστολής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Φερχόφστατ, που είσαστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και εμείς σας ευχόμαστε να τα καταφέρετε σε αυτές τις δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις και οπωσδήποτε ευελπιστώ ότι δεν, ήταν αυτή η, δεν θα είναι αυτή η τελευταία φορά που θα σας συναντήσουμε και θα σας ακούσουμε εδώ. Uh, dear members, we still... Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε δύο ακόμα σημεία στην ημερήσια διάταξη πριν τη διακοπή. Ελπίζω να μην έχετε εξαντληθεί τόσο πολύ ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε. So if you allow me... Αν μου επιτρέπετε λοιπόν... Συνεχίζουμε με το σημείο 13. προστασία των επιχειρηματικών μυστικών. Τον λόγο έχει η κυρία Λεγκρίπ. Παρακαλώ ησυχία στην αίθουσα Παρακαλώ ησυχία, ηρεμία Very Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήρθα εδώ ενώπιόν σα ε, σήμερα το πρωί έτσι ώστε να σας ε, αναφέρω το στάδιο στο οποίο έχουμε φτάσει όσον αφορά τον τριμερή διάλογο εντός εισαγωγικών σύμφωνα με την εντολή την οποία είχα όσον αφορά τα εμπορικά απόρριτα. Θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει συνάντηση τρι, τριμερούς διαλόγου ε, προκεχωρημένη της νυχτός και επομένως είμαστε όλοι σε πολύ καλή κατάσταση και καταφέραμε ε, ε, να είμαστε ιδιαίτερος ε, ε, σε, σε πολύ καλή φόρμα και ξύπνοι την ώρα που κάναμε τον τριμερή διάλογο. Στις 16 Ιουνίου του 2015 λοιπόν έγινε ψηφοφορία και σχετική εντολή. Έκτοτε είχαμε δύο συνεδριάσεις, μία το Σεπτέμβριο κράτησε δύο ώρες, ήταν μια πρώτη την έτσι, ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, και ήρθαμε σε επαφή με τους ΔΕ και η δεύτερη στις 27 Οκτωβρίου στη διάρκεια της Ολομελίας στο Στρασβούργο. Ε, πρόκειται για μία συνεδρίαση η οποία κράτησε δύο ώρες ε, και η οποία μας έδωσε την ε, δυνατότητα να ε, δούμε ποια ήταν ακριβώς τα σημεία τα οποία παρουσίαζαν μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί στις 27 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο καταφέραμε να κάνουμε έναν κατάλογο μέσω ανταλλαγής απόψεων των τριών σε έναν ειλικρινή και χωρίς υποχωρήσεις διάλογο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ε, καταλήξαμε λέω σε ένα κατάλογο των προβλημάτων χωρίς όμως να έχουμε προχωρήσει σε καμία ε, πρόοδο ας πούμε, χωρίς να έχουμε μπει δηλαδή στην ουσία ε, του πράγματος. Είδαμε πάντως ποια είναι τα ισχυρά σημεία, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές των θέσεων των μεν και των δε. Η σκιώδη συζητής και εγώ η ίδια είχα τη δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις μας στο Συμβούλιο. Επίσης ε, ε, το Συμβούλιο ακούσαμε ε, να μας λέει ότι εξ ονόματος του Συμβουλίου μπορούσε να πει ότι το Συμβούλιο θέλει να συναντήσει τις ε, θέσεις ε, του Κοινοβουλίου και εμείς σημειώσαμε λοιπόν αυτή την καλή θέληση που εξέφρασε το Συμβούλιο. Είναι γεγονός ότι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ε, συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου το Συμβούλιο είχε κάνει και μια συνεδρίαση κορεπέρ οπότε είχε συζητήσει κάποια ζητήματα τα οποία μπορούσαν να αφήνουν κάποια ευελιξία ή κάποιο ε, περιθώριο ελιγμών. Ε, μετά από την ε, συνάντηση της 27ης Οκτωβρίου, το Συμβούλιο αλλά και η Κομισιόν όσον αφορά ορισμένα θέματα μας γνωστοποίησαν ότι θα υποβάλουν νέες προτάσεις επί σειρά θεμάτων, δηλαδή θα μας κάνουν ε, νέες διατυπώσεις κειμένου ε, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι πιο κοντά στις δικές μας θέσεις κυρίως όσον αφορά πολλά ουσιώδη ζητήματα τα οποία υποβάλαμε. Το θέμα της διαφάνειας της πληροφόρησης ας πούμε καθώς επίσης ε, και της πλήρου και άμεσης ε, ε, ελευθερίας έκφρασης και δράσης, ε, το θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων και το γεγονός δηλαδή ότι σε περίπτωση προστασίας κάποιου απορρίτου, εμπορικού απορρίτου δεν θα μπορούσε να παρεμποδιστεί η ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων και η προώθηση της επαγγελματικής τους διαδρομής και καριέρας. Επίσης, ε, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ θετικό αυτό το, το βήμα από πλευρά της Προεδρίας γιατί δείχνει ότι πραγματικά έχουν την διάθεση και τη θέληση να προχωρήσουν στι διαπραγματεύσεις κάνοντάς μας ε, ε, συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης, τις οποίες λάβαμε πριν από μερικές ε, μέρες, στην αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα, στα πλαίσια της τεχνικής συνάντησης, που έδωσε τη δυνατότητα στο επίπεδο το οποίο συνεχίζουμε να ονομάζουμε τεχνικό, να μελετήσουν αυτές τις συγκεκριμένες διατυπώσεις, τις επαναδιατυπώσεις του άρθρου 1, του άρθρου 2, ε, μιας ε, ε, επαναδιάρθρωσης επίσης του άρθρου 1 σε σχέση με το άρθρο 4, γιατί θυμίζω ότι εμείς είχαμε στην έκθεση τροποποιήσει την διάρθρωση των άρθρων. Κυρίως είχαμε μεγαλώσει το άρθρο 1 του σχεδίου οδηγίας, εντάσσοντας σε αυτό το άρθρο 1 μία σειρά στοιχείων και σκέψεων, όσον αφορά τα θέματα, τα διακυβεύματα και τους ε, τομείς επί των οποίων η παρούσα οδηγία θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο. Ξεκίνησε λοιπόν μια ε, πραγματική ουσιαστική συζήτηση με το Συμβούλιο όσον αφορά την επαναδιατύπωση και τον συσχετισμό των άρθρων, κυρίως ε, συσχετισμός άρθρου 1 και άρθρου 4 όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις Ε, γιατί ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει σαφής, σαφής αναφορά στους whistleblowers, στα μέσα ενημέρωσης και κυρίως στους λεγόμενους δημοσιογράφους ερεύνης και επ' αυτών λέω έχουν ε, υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις ε, επαναδιατύπωσης ε, τις οποίες θα πρέπει να διαβάσουμε, να αναλύσουμε, να ξεψαχνίσουμε αν μου επιτρέπετε την έκφραση έτσι ώστε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Εδώ βρισκόμαστε. Έχουμε φτάσει στα πρώτα άρθρα τα οποία εμείς τα είχαμε δουλέψει όπως σας έχω πει επανειλημμένα ε, και επομένως κυρίως τη διασύνδεση αυτή του άρθρου 1 με το άρθρο 4. Επ' αυτού λοιπόν έχουμε καινούριε προτάσεις διατύπωσης ε, τις οποίες μας έχει υποβάλει το Συμβούλιο και... Ε, Οπωσδήποτε ε, σύντομα η ε, η ομοδιαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου ε, θα, θα καταρτήσει έναν χάρτη πορείας. Ε, πολύ σύντομα θα συναντηθούμε έτσι ώστε να συζητήσουμε αυτές τις νέες προτάσεις διατύπωσης που έχει υποβάλει το Συμβούλιο έτσι ώστε να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η, ε, η απάντηση βάσει επιχειρημάτων που θα μπορούσαμε να δώσουμε στο Συμβούλιο και που θα μπορούσε να ενταχθεί στην δέσμη διαπραγματεύσεων και τον τρόπο γενικά με τον οποίο ε, θα αποφασίσουμε να συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις. Ε, σκεφτόμαστε να κάνουμε μια νέα συνάντηση τριμερούς διαλόγου περί τα τέλη Νοεμβρίου με την ευκαιρία της επόμενης Συνόδου Ολομελίας. Επομένως, σε αυτή τη φάση. Καμία ουσιαστική πρόοδος, καμία ε, απτή πρόοδος. Ε, απλώς καταγράφουμε την βούληση του Συμβουλίου ε, να ακολουθήσει μια συνεδρική οδό με την έννοια να κάνει κάποιες κινήσεις ε, καλής θελήσεως τις οποίες ε, καταγράφουμε γιατί αφορούν ε, πολύ συγκεκριμένα σημεία και σημεία ε, στα οποία αποδίδουμε μεγάλη σημασία. θα συναντηθούμε με τους σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε συγκεκριμένα να διαβάσουμε και να συζητήσουμε και να μελετήσουμε αυτές τις νέες προτάσεις διατύπωσης του Συμβουλίου. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. γιατί υπάρχουν και κάποια στοιχεία της διαπραγμάτευσης που και δύσκολα είναι και επίπονα, αλλά σε αυτή τη φάση μπορούμε να πούμε ότι επί ορισμένων σημείων και επί ορισμένων θεμάτων οι προτάσεις επαναδιατύπωσης είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσες. Κυρίως το κύριο μέλημά μας, ε, δηλαδή ε, να μην εμποδιστεί με κανένα τρόπο η πλήρης ε, επαγγελματική κινητικότητα ε, των υπαλλήλων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ήθελα να σας πω. Οι σκιώδεις θα ξανασυναντηθούν έστω και αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες έτσι να βρούμε την ημερομηνία που θα βολεύει όλους. Έναν επόμενο τριμερή διάλογο, όπως σας είχα πει, τέλη Νοεμβρίου και πάντως ε, το μήνυμα είναι ότι βλέπουμε μια καλή επικοδομητική δυναμική, βλέπουμε ε, μια διάθεση του Συμβουλίου έτσι να δείξει καλή θέληση. Ε, υπάρχει λοιπόν μια επικοδομητική διάθεση, πράγμα που σημαίνει ότι βήμα-βήμα μπορούμε να χτίσουμε κάτι λογικό και ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο το λόγο και επομένω μπορούμε να ζητήσουμε από τον κύριο Κοφεράτη ε, να μας πει ε, στα έξι λεπτά που μας μένουν νομίζετε ότι μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε την έκθεσή σας. Α, φαίνεται πως ναι. Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, για το σημείο 14. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, λέει ο κ. Κοφεράτη. Και γιατί ο τριμερής διάλογος ε, ε, ήταν μόνο ένας σχετικά με το, την οδηγία για τα δικαιώματα ε, των ε, μετόχων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, προεδρία σας και για τη βοήθεια που δώσατε σε αυτήν την περίπτωση. Σε γενικές γραμμές μελετήσαμε τα κύρια στοιχεία της οδηγίας σχετικά με την ενεργή συμμετοχή των μετόχων, σχετικά με την διαφάνεια, σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας και την ψήφο κτλ. Εμείς ε, βρήκαμε κάποια στοιχεία σύγκλησης αλλά και ισχυρότατα σημεία απόκλησης. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να προχωρήσω ως εξής. Να προχωρήσουμε λοιπόν με τεχνικές συναντήσεις, μία αύριο, μία στις 16 Νοεμβρίου και μία άλλη τρίτη στις 30 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να γίνει μία προσπάθεια επί των γραπτών κειμένων να ε, δούμε τα σημεία ε, σύγκλησης. Πάντως έχουμε προκαθορίσει μία αρχή ότι το συμπέρασμα όταν και εφόσον υπάρχει θα πρέπει να αφορά όλα τα ε, ε, θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Ε, δηλαδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε επιμέρους λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα και να διχάσουν και επί θεμάτων τα οποία μεταξύ τους έχουν μεγάλη συνάφεια. Επομένως μπορούμε να αξιολογήσουμε θετικά ένα καλό κλίμα που διαπιστώσαμε στον πρώτο τριμερή διάλογο. Δεν σας κρύβω ότι ε, πέραν της εγκαρδιότητος εξεφράστησαν και ε, ε, απόψεις εξαιρετικά διεστάμενες όσον αφορά ορισμένα ζητήματα τα οποία εν μέρει έχω αναφέρει κυρίως εκ μέρους του Συμβουλίου. Μετά τις τεχνικές ε, ε, συνεδριάσεις ε, και υπό το φως των, της έκβασης αυτών των τεχνικών συνεδριάσεων θα μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα συνάντηση και βεβαίως μετά από συζήτηση και με τους χιώδης ηγητές θα είμαι σε θέση να σας δώσω μια αξιολόγηση πιο συγκεκριμένη και απτή γιατί σήμερα δεν είμαι σε θέση να κάνω κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ξέχασα, γιατί δεν είχα όλη την, ε, ε, ε, την ημερήσια διάταξη. Έχουμε τον κύριο Ζαμπάφκη. Μήπως οι διερμηνείς μπορούμε να μας δώσουν μερικά λεπτά έτσι ώστε ο κύριος Ζαμπάσκη να κάνει την παρουσίασή του. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε θα μιλήσει τη γλώσσα μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, πριν μπω στις λεπτομέρειες της πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας πω το χρονοδιάγραμμα. 3 Δεκεμβρίου το σχέδιο θα παρουσιαστεί το σχέδιο γνωμοδότησης 9 Δεκεμβρίου προθεσμία για τροπολογίες ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότησης 28 Ιανουαρίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 30 Νοεμβρίου και 1 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί η έκθεση και 11 Νοεμβρίου προθεσμία για τροπολογίες ψηφοφορία στα μέσα Φεβρουαρίου Ο κανονισμός αυτός τροποποιεί τον κανονισμό του 95 ο προηγούμενος ο κανονισμός έχει τροποποιηθεί ήδη δύο φορές αλλά οι τροπολογίες αυτές ε, δεν αφορούσαν ε, τη μορφή του αυτοκόλλητου της ε, βίζας της θεώρησης γιατί υπήρχαν διάφορα πλαστά τέτοια αυτοκόλλητα οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Συμφωνώ πλήρως λοιπόν με τις προτάσεις της Κομισιόν για το ότι πρέπει η πλαστογραφία να γίνει και θα γίνει σχεδόν αδύνατη. Η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ελπίζω να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι. Αν με έχουν ενημερώσει τώρα σωστά, υπάρχει ένας εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν και μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ σύντομα κύριε Πρόεδρε ξέρω πως ε, η πρόταση έχει στήριξη γιατί υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις ε, πλαστογραφίας οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Μάλιστα, θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Οπότε τελειώσαμε στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές ε, και συνεχίζουμε στις 3 ε, με την μήνυα ακρόαση.